Good morning everybody. Please take your seats. Καθίστε παρακαλώ. I know it's very emotional to be together again. Ξέρω ότι είναι πολύ συγκινητικό που ξαναβρισκόμαστε μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. But anyway, we... Πάντως, έχουμε σοβαρή δουλειά να κάνουμε σήμερα. Καθίστε παρακαλώ. Ελπίζω, ξεκινώ μάλλον την συνεδρίαση της έκτακτης αυτής ε, συνάντησης της Επιτροπής Ανάπτυξης. Είστε ενημερωμένοι για την ημερήσια διάταξη. Έχετε κάποιες προτάσεις. Δεκτή λοιπόν. Ανακοινώσεις της Προέδρου, μία μόνη ανακοίνωση. Να σας καλωσορίσω. Ελπίζω να είναι επιτυχής η συνάντησή μας. Ελπίζω να έχετε όλοι καλή υγεία. Είναι μεγάλη χαρά που συνεργαζόμαστε στην Επιτροπή Ρέγγι. Και θα συνεχίσουμε με το ίδιο πνεύμα. Αυτό είχα να πω σήμερα. Το τέταρτο σημείο είναι το βασικό σημείο βέβαια. Όλοι γνωρίζετε τις οικονομικές δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζει η Ελλάδα και τη συμφωνία η οποία υπήρξε στις 13 και 14 Ιουλίου για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για περαιτέρω οικονομική βοήθεια προς την Ελλάδα. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε μια νομοθετική πρόταση για την αναθεώρηση του κανονισμού κοινών διατάξεων για τη λήψη έκτακτων μέτρων για βοήθεια προς την Ελλάδα. Ε, η Επίτροπος ε, μας ζήτησε να παρουσιάσει τις προτάσεις της αυτές σήμερα. Χαιρετίζω την Επίτροπο, την ευχαριστώ για την παρουσία της. Η Επίτροπος Κρέτσου θα παρουσιάσει τις προτάσεις της. Θα πρέπει όμως να πω κάποια πράγματα σχετικά με την διαδικασία η οποία θα ακολουθηθεί στο Κοινοβούλιο. Η επίσημη έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας θα γίνει όταν λάβει επίσημα, μάλλον ανακοινώσει επίσημα στην Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου την παραλαβή της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ορίσει ως υπεύθυνη επιτροπή την δική μας επιτροπή και επίσης θα ζητήσει γνωμοδοτήσεις από την Επιτροπή Απασχόλησης, Γεωργίας και Αλίας. Ταυτόχρονα θα υπάρξει δυνατότητα διαβούλευσης για την Επιτροπή των Περιφερειών και για την Κοινωνική και Οικονομική Επιτροπή. Οι γνωμοδοτήσεις τους θα πρέπει να μας δοθούν μέχρι το τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου είναι κάτι το οποίο έχει ήδη γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης ε, σε επίπεδο πρωτοβουλειών προς το παρόν με τα δύο αυτά σώματα. Το Συμβούλιο έχει ήδη ξεκινήσει τις εργασίες του. Η Ομάδα Εργασίας Διαφθορωτικών Δράσεων ε, συνεδρίασε στις 24 Ιουλίου και θα συναντηθεί εκ νέου αύριο και μετά στις 11 Σεπτεμβρίου. Οι συντονιστές συναντήθηκαν νωρίτερα σήμερα για να συζητήσουν τις διάφορες διαδικαστικές διαδικασίες οι οποίες υπάρχουν για την Επιτροπή Ανάπτυξης. Στις συζητήσεις μας σήμερα, πριν ξεκινήσουν, θα αναφερθώ και στα συμπεράσματα αυτών των συναντήσεων. Θέλω πάντως να καλωσορίσω την αρμόδια Επίτροπο για την Περιφερειακή Πολιτική. Θα μας παρουσιάσει την πρότασή της. Μετά την παρουσίασή της, στα μέλη, για τα σχόλιά τους και τις ερωτήσεις τους ξεκινώντας από τους συντονιστές. Όλοι επιθυμούμε να έχουμε σωστά οργανωμένες συνεδριάσεις των Επιτροπών μας και γι' αυτό θα περιορίσω τα σχόλια των μελών χρονικά έτσι ώστε όλοι όσοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στη συνάντηση και στη συζήτηση να έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Έχετε το λόγο. Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, συνάδελφοι, καλημέρα σας. Είναι μεγάλη χαρά για μένα που επανέρχομαι εδώ ανάμεσά σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω που αποφασίσατε να κάνετε αυτή την έκτακτη συνεδρίαση για να συζητήσετε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροπολόγηση των κανονισμών κοινών διατάξεων για την Ελλάδα σχετικά με τα ειδικά μέτρα για την Ελλάδα. Είναι ένα έκτακτο μέτρο αν θέλετε για να ε, αντιμετωπιστεί μια έκτακτη κατάσταση στην Ελλάδα. Και ο παράγων εδώ ο οποίος θα είναι καθοριστικός για την επιτυχία αυτών των μέτρων θα είναι ο χρόνος. Γνωρίζουμε την κατάσταση στην Ελλάδα, δραματική η κατάσταση στην Ελλάδα. Τα είχαμε συζητήσει και λίγο πριν το καλοκαίρι σχετικά με την επίσκεψη την οποία θα έκανα σε διάφορες ελληνικές περιφέρειες Εκεί εντυπωσιάστηκα από το θάρρος και την αφοσίωση των ανθρώπων τους οποίους συνάντησα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι αξίζει της υποστήριξής μας η Ελλάδα. Ως εκ τούτου λοιπόν έχει μεγάλη σημασία να καταλήξουμε σε μια συμφωνία επί της προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροπολόγηση του κανονισμού και των κοινών διατάξεων. Το ταχύτερο δυνατόν. Είναι μια πολύ σοβαρή κρίση και έχει συνέπειες ε, σε επίπεδο οικονομικών ε, πολιτικών και οδήγησε και στην κρίση ρευστότητας της Ελλάδας. Έχει τεράστιες προκλήσεις για την μεταρρύθμιση της οικονομίας της και να περάσει στο δρόμο της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στήριξε την Ελλάδα και σε επίπεδο τεχνικής βοήθειας και σε επίπεδο οικονομικής βοήθειας. Στις 15 Ιουλίου εκδώσαμε μια ανακοίνωση λέγοντας μια νέα αρχή για την ανάπτυξη και τη δουλειά και την απασχόληση στην Ελλάδα. Λέμε εκεί ότι υπάρχουν ικανοποιητικά μέσα από πλευρά του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να ξεκινήσει εκ νέου η ευρωπαϊκή οικονομία. Η συμφωνία της 12ης Ιουλίου και οι λεπτομέρειες του τριμερούς προγράμματος στα πλαίσια του ESM έχουν ε, σαν στόχο την δημοσιονομική ισορροπία και την δημιουργία ενός σταθερού κλίματος επενδυτικού έτσι ώστε να ξεκινήσει εκ νέου ε, να λειτουργεί η ελληνική οικονομία. Είναι κρίσιμο η Ελλάδα βέβαια να εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις αυτές που θα δώσουν την δυνατότητα στη χώρα να χρησιμοποιήσει 86 δις ευρώ σε δάνεια τα επόμενα τρία χρόνια. Αυτό θα βοηθήσει και τις επενδύσεις στον ιδιωτικό τομέα και θα βοηθήσουν στην βιωσιμότητα της ελληνικής οικονομίας. Α, όλα αυτά τα μέτρα λοιπόν είναι απαραίτητα αλλά δεν είναι από μόνα τους επαρκή, πρέπει να προκαλέσουν και ιδιωτικές επενδύσεις. Το θέμα δεν είναι να δαπανηθούν οι πιστώσεις αυτές, το θέμα είναι να δαπανηθούν σωστά και οι ευρωπαϊκές πιστώσεις εδώ θα παίξουν ένα σημαντικό ρόλο. Είναι διαθέσιμα τα ποσά, είναι καθορισμένα τα ποσά, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν το ταχύτερο δυνατόν. Στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 17η Ιουλίου υιοθέτησε μία πρόταση για την τροπολόγηση του κανονισμού κοινών διατάξεων έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά προβλήματα ρευστότητας που παρεμποδίζουν τη σωστή εφαρμογή των μέτρων που ακολουθούν τις ευρωπαϊκές πιστώσεις προς την Ελλάδα. Να υπάρξει... Ε, holding back supported by... Να υπάρξει εκ των προτέρων καταβολή των πιστώσεων, το λεγόμενο front loading, όπως επίσης και μέτρα για τη σωστή κατάληξη του προγράμματος 2007-2013. Τι σημαίνουν όλα αυτά. 2014-2013 η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η αύξηση της προχρηματοδότησης κατά 7% για το ERDF και για τα Ταμεία Συνοχής όπως επίσης και για το Ταμείο ε, για την Αλία αυτή η έκτακτη προχρηματοδότηση θα καταστήσει σε επίπεδο διετίας ένα δις επιπλέον διαθέσιμο για το 2015 και το 2016. Αυτό θα επιτρέψει να ξεκινήσουν περισσότερα προγράμματα και με μεγαλύτερη ταχύτητα, υψηλότερη ταχύτητα. Οι συμπληρωματικές ανάγκες προχρηματοδότησης θα συμπληρωθούν με τις πληρωμές στο τέλος του 2013. Για την περίοδο 2007-2013 έχουμε ε, προτείνει εμείς να δοθούν τα τελευταία εναπομείναντα 5% των πληρωμών που έχουν ε, κρατηθεί θα έλεγε κανείς μέχρι ότου κλείσει επίσημα το πρόγραμμα. Προτείνουμε επίσης και εθνική συγχρηματοδότηση μηδενική μέσω δηλαδή ε, συγχρηματοδότησης από πλευράς μας κατά 100%. 500 περίπου εκατομμύρια αυτό σημαίνει το 2015 και ένα αντίστοιχο πάλι 500 εκατομμυρίων το 2016. Αυτό θα ελαφρύνει τις πιέσεις σε δημοσιονομικό επίπεδο στην Ελλάδα και συνιστά μια ουσιαστική αύξηση των διαθεσίμων πιστώσεων. Δηλαδή θα διατεθούν με λίγα λόγια τα ποσά τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν κρατηθεί λόγω της έλλειψης συγχρηματοδότησης από την εθνική πλευρά, από την ελληνική πλευρά. Τα μέτρα αυτά λοιπόν θα επιτρέψουν τη σωστή και πλήρη εφαρμογή ε, όλων των ρυθμίσεων 2007-2013. Είναι σαφές βέβαια τα χρήματα αυτά να φτάσουν σε αυτούς οι οποίοι τα έχουν ανάγκη το ταχύτερο δυνατόν και να υπάρξει χρηστή ε, οικονομική διαχείριση αυτών των ποστών. Και εδώ τίθεται και το θέμα του CPR και ζητάτε να δημιουργηθεί το λεγόμενο ring fencing, ένας αμυντικός μηχανισμός δηλαδή, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν τα ποσά αυτά μόνο για πληρωμές προς τους οποίους κατευθύνονται και είχαν προβλεφθεί. Στις ε, αρχές Αυγούστου ε, ελήφθησαν αυτές οι αποφάσεις και ζητήθηκε από την Ελλάδα να αναφέρεται τακτικά για τις εφαρμογές του μέτρου αυτού μέχρι το τέλος του 2016 και να υπάρξει και η τελική έκθεση για την περίοδο 2007-2013 σε επίπεδο δημοσιονομικών βαρών. Τα μέτρα αυτά δεν δημιουργούν προβλήματα σε επίπεδο MFF και σε επίπεδο πληρωμών και σε επίπεδο υποχρεώσεων. Θα οδηγηθούμε σε ένα περιορισμένο front loading το οποίο είναι δημοσιονομικά ουδέτερο για το MFF. Αυτό το front loading για το 2015 θα καλυφθεί από τα ποσά τα οποία έχουν προβλεφθεί για την περίοδο 2014-2020. Για το 2016 τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογήσει τις προβλέψεις της αναθεωρημένες των κρατών μελών και την δημοσιονομική κατάσταση σε επίπεδο εφαρμογής. Μετά από την αξιολόγηση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει τις ρυθμίσεις της για το 2016 αν χρειαστεί. Νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε λοιπόν ότι τα μέτρα αυτά θα βοηθήσουν ιδιαιτέρως, θα είναι ευεργετικά για την ελληνική οικονομία. Οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνεργάζονται στενά με τις ελληνικές αρχές οι τεχνικές συνεδριάσεις και οι αποστολές ad hoc στην Ελλάδα οργανώνονται συνεχώς και θα υπάρξει περαιτέρω έλεγχος σε σχέση ε, με τις ε, αναφορές τις οποίες θα πρέπει να κάνουν οι ελληνικές αρχές. Οι επενδύσεις αυτές θα πρέπει να στοχεύουν στις πραγματικές ανάγκες και να επηρεάσουν με ουσιαστικό τρόπο την ελληνική οικονομία. Ένα παράδειγμα ίσως να σας δώσω του τι εννοεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργαζόμαστε με την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στα πλαίσια της προπαρασκευαστικής δράσης για την εκλέπτυνση των στόχων της στρατηγικής σε τομείς υψηλής δυνατότητας για την αύξηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στην περιοχή αυτή. Οι πιστώσεις μας έχουν βοηθήσει πολύ στην ενίσχυση της ε, ελληνικής οικονομίας, έχουν βοηθήσει πολύ την οικονομική και την κοινωνική συνοχή. Τώρα που η Ελλάδα αντιμετωπίζει περισσότερα προβλήματα έχει μεγάλη σημασία να υιοθετηθεί από εσά η πρότασή μα το ταχύτερο δυνατόν για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα ρευστότητα που παρεμποδίζουν τη σωστή χρήση των κοινωνικών κοινοτικών πιστώσεων στην Ελλάδα. Φυσικά το Συμβούλιο και εσείς είσαστε υπεύθυνοι για την υιοθέτηση αυτής της νομοθετικής τροποποίησης. Νομίζω ότι στην παρούσα φάση ο χρόνος μετράει για να πετύχει η προσπάθεια αυτή. έτσι ώστε να κλείσει το θέμα των υπόλοιπων ποσών από το 2007-2013 και να απορροφηθούν οι πιστώσεις αυτές από την οικονομία που τα έχει ανάγκη. Ελπίζω λοιπόν το ταχύτερο δυνατόν να γίνει δεκτή η νομοθετική πρόταση και στηρίζομαι στην δική σας προσπάθεια. Είμαι στη διάθεσή σας να ακούσω τα σχόλιά σας αν έχετε ερωτήσεις. Και ελπίζω αυτό το τελευταίο τμήμα του χρόνου να χαρακτηριστεί από σωστή συνεργασία και εντατική ανάμεσα στην Επιτροπή και εσάς. Ευχαριστώ Επίτροπε. Θα ξεκινήσω με τους συντονιστές. Τρία λεπτά ο κάθε συντονιστής. Τρία λεπτά. Βανίστελ Ρόι. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτήν την συνεδρίαση και ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση την κυρία Κρέτσου. Νομίζω πως γνωρίζουμε όλη την ε, κατάσταση που στην Ελλάδα και γνωρίζουμε βέβαια και τη θέση του Συμβουλίου. Αλλά θα πρέπει να δούμε και ποια είναι η δική μας, ε, ε, ο δικός μας όλος ως Επιτροπή Ρέτζη. Είναι να προετοιμάσουμε δηλαδή το τι θα συζητηθεί σε επίπεδο ολομέλειας. Και εκείνο που είναι σημαντικό για μένα είναι να μην δημιουργήσουμε προβλήματα στην στάση που θα θελήσει να υιοθετήσει το Κοινοβούλιο. Και βάσει την ποιότητα των δεδομένων που λάβαμε, θα αποφασίσουμε. Δηλαδή, μας είπατε ότι αν καταργήσουμε τη συγχρηματοδότηση, δεν θα υπάρξει μείωση των επενδύσεων από την ελληνική πλευρά. Ε, δηλαδή στην πραγματικότητα η ε, χρηματοδότηση είναι 105% γιατί η συγχρηματοδότηση ελληνική θα παραμείνει μέσα στα περιφερειακά προγράμματα και εμείς αυξάνουμε το ποσοστό συγχρηματοδότηση από την πλευρά μας στο 100%. Έχουμε λοιπόν μία σειρά από ερωτήσει και έκανα και το Συμβούλιο ερωτήσεις γιατί προετοιμάζεται ακόμα και απάντησε σε όλα αυτά τα ερωτήματα η Επιτροπή. Οπότε θα θέλαμε και εμεί να λάβουμε και εμεί τι απαντήσει μα. Μέσα δηλαδή στην επόμενη εβδομάδα θα πρέπει να έχουμε μια διαδικασία που να μα επιτρέψει να θέσουμε ερωτήματα στην Επιτροπή και να λάβουμε, να λάβουμε αυτές τις απαντήσεις γραπτώς. Και αυτό το λέω γιατί φοβάμαι ότι θα συμβεί το εξή. Είναι πολύ ωραία βέβαια όλα το ότι μπορούμε να φτάσουμε σε μια πολιτική συνένεση ώστε να διαφυλάξουμε ε, τα συμφέροντα της Ελλάδας προς το παρόν να το πω και αυτό, ελπίζοντα ότι όλα αυτά θα λειτουργήσουν, αλλά εν πάση περιπτώσει στο τέλο ε, μπορεί το πρόβλημα να είναι ότι αυτά τα χρήματα τα οποία θα επενδύσουμε εμεί να πάνε κατευθείαν στι τράπεζε και να μην απορροφηθούν από την ελληνική οικονομία. Ε, Εμεί θέλουμε πραγματικά λοιπόν να έχουμε έναν προπολογισμό που θα είναι επενδυτικό για την Ελλάδα. Οπότε θέλουμε να ξέρουμε ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι, ποιοι θα λάβουν αυτά τα χρήματα. Και όπω είπατε και εσεί, είναι σημαντικό να λάβουν αυτά τα χρήματα οι δικαιούχοι. Κατά συνέπεια, έχουμε ερωτήματα εμεί ακόμα, ε, τα, τα μέλη τη ομάδα μου έχουν ε, διάφορε ερωτήσει και μου είπαν ε, Μόλι γύρισα από τι διακοπέ μου τα μέλη τη πολιτική μου ομάδα ότι θα, θέλαν, θα ήθελαν να έχουν το δικαίωμα να ε, καθέσουν τροπολογίε. Γιατί ε, μεταξύ άλλων δεν ξέρουμε ε, εάν το Συμβούλιο θα καταθέσει τροπολογίε. Πώ λοιπόν, γιατί να εκχωρήσουμε αν θέλετε, να μην αξιοποιήσουμε το δικαίωμα μα, να βάλουμε εμεί ε, τροπολογίε. Δεν θα πρέπει όπω ε, και τα άλλα θεσμικά όργανα να έχουμε και εμεί τη δυνατότητα να υποβάλουμε τροπολογίε και να μην περιθωριοποιηθούμε ας έχουμε τουλάχιστον μια γραπτή διαδικασία για να προετοιμάζουμε ε, τις ε, συνεδριάσεις μας και να μην λαμβάνουμε έτσι από το πουθενά κάποιες ε, πληροφορίες άμεσα. Συνοψίζοντας λοιπόν, η προτίμηση του δικού μα της παιδικής μας πολιτικής ομάδας είναι να έχουμε μια ε, διαδικασία με υπόβολο τροπολογία. Ε, μια κανονική διαδικασία. Και μάλιστα εμεί είχαμε προτείνει να δίνουν δύο εξαιρετικέ συνεδριάσει ε, τη ΡΕΤΖΙ, ώστε να μην έχουμε κολλήματα για την άσκηση των δικαιωμάτων από πλευρά των δικών μα μελών. Δεν πρέπει να είμαστε ευέλικτοι. Η Επιτροπή των Περιφερειών έχει το δικαίωμα να περιμένει μήνε μέχρι να προετοιμάσει τη γνωμοδότησή του. Εμεί δεν έχουμε αυτό το δικαίωμα ω Κοινοβούλιο, να δώσουμε δύο-τρει μήνε στον εαυτό μα. Δεν πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να δρούμε και να μην δημιουργούμε προβλήματα στην των δικαιωμάτων από πλευρά των μελών του ε, Κοινοβουλίου. Αν το κάνουμε αυτό θα έχουμε αποτύχει στα καθήκοντά μας. Οπότε ε, αυτά από τη δική μας πλευρά και ε, πραγματικά επαφήμαι σε εσάς πρώτα για να έχουμε μια σωστή συζήτηση με τους συναδέλφους. Και μάλιστα ε, επί τη βάση γραπτών κειμένων, όχι απλά έτσι στον αέρα. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. κύριε Βανίστερο, θα πρέπει να σας απαντήσω. Δεν έγινε συνάντηση, συνεδρίαση της Επιτροπής μας τον Απρίλιο γιατί βρισκόμασταν και πάρα πολύ μακριά από τη σημερινή κατάσταση και από τα ζητήματα που συζητάμε σήμερα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε όλοι μαζί, ούτω ώστε να βελτιώσουμε βέβαια και τον τρόπο που λειτουργεί η Επιτροπή μα στο πλαίσιο πάντα βέβαια των εργασιών του συνόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί όλε οι επιτροπές ε, κοινοβουλευτικέ αντιμετωπίζουν προβλήματα στο πλαίσιο τη άσκηση, δηλαδή εντολή εντολής τους, ε, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Α μην μπλέκουμε τώρα αυτό το θέμα με το ζήτημα που συζητούμε. Ας εστιάσουμε λοιπόν στο ζήτημα που θέλουμε να επιλύσουμε σήμερα και το οποίο θέλουμε να συζητήσουμε. Κυρία Κρέλ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε ενώπιον μιας ε, εξαιρετικής ε, κατάστασης ε, για την Ελλάδα και θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, Επίτροπο για το γεγονός ότι μετά από διάσκεψη κορυφής στις 12 και 13 Ιουλίου αντέδρασε πάρα πολύ γρήγορα και υπέβαλε μία πρόταση εδώ επιτάπητος επί της οποίας θα μπορούσαμε κατά δική μου άποψη να αποφασίσουμε ήδη σήμερα γιατί δεν αντιλαμβάνομαι πώς μπορούν να υπάρχουν αντιρρήσεις αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση όμως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι οπωσδήποτε υποχρεωμένο. Έχει δηλαδή αυτή την ηθική υποχρέωση να βοηθήσει το ταχύτερο δυνατό ε, τον ελληνικό λαό. Νομίζω πως έχουμε συζητήσει ξανά και ξανά και εδώ σε αυτή την Επιτροπή το τι χρειάζεται η Ελλάδα για να προχωρήσει. Και πάντα η δική μας άποψη ήταν ότι θα πρέπει να επενδύσουμε στην Ελλάδα ούτως ώστε να σταθεί και πάλι στα πόδια της ελληνική οικονομία και έτσι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους εκεί, να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, να παράσχουμε ε, κοινωνική ασφαλεία. Οπότε πώς μπορεί κάποιος εδώ, μέλος του Κοινοβουλίου, να αντιταχθεί σε, στη, στην προτινόμενη απλουστευμένη διαδικασία και, ε, ε, στο να υλοποιηθεί δηλαδή γρήγορα ε, το αποτέλεσμα της τα κράτη-μέλη έχουν ε, ε, κινηθεί με μια ανοιχτή ε, διαδικασία, διαφανή διαδικασία, μπορεί κανείς δηλαδή να δει όλα τα έγγραφα, οπότε δεν αντιλαμβάνω από πού μπορούν να προκύψουν περαιτέρω ερωτήματα πέρα δηλαδή από αυτήν την προτινόμενη τροποποίηση των σχετικών άρθρων του κανονισμού περί κοινών διατάξεων. Δεν λέμε ότι κανείς πρέπει να καταβάλει κάποιο ποσό παραπάνω, απλά λέμε όλα τα προγράμματα προσπαθούμε να τα οριστικοποιήσουμε το ταχύτερο δυνατό ώστε να έρθουν γρήγορα σε αυτή τη χώρα οι επενδύσει ε, που χρειάζεται. Δηλαδή, οι επενδύσει οι οποίε ήδη έχουν αποφασιστεί ότι θα εστρέψουν στην Ελλάδα, αποφασίζουμε τώρα να ελοποιηθούν το ταχύτερο δυνατόν. Να εστρέψουμε στην Ελλάδα το ταχύτερο δυνατό. Οπότε, η δική μου πολιτική ομάδα δεν θέλει να ξεκινήσει τώρα μια συζήτηση ε, κατά πόσο θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τώρα ε, το δικαίωμά μα ή όχι, το να ασχοληθούμε με ένα τέτοιο ζήτημα μέσω τη ε, ε, διαδικασία. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια εξαιρετική περίπτωση περίπτωση, οπότε θα πρέπει να αξιοποιήσουμε και εξαιρετικά μέτρα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει πραγματικά να ακολουθήσουμε μια ταχύτατη διαδικασία και να απευθύνουμε μια έκκληση στο Συμβούλιο να πράξει το ίδιο. Έχουμε δηλαδή επανειλημμένα μια κατάσταση όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι διατεθειμένο να δράσει ταχύτατα και από την άλλη πλευρά το Συμβούλιο να δημιουργεί καθυστερήσει. Οπότε σε κάθε περίπτωση και τα δύο αυτά θεσμικά όργανα ε, θα πρέπει να πιεστούν όσο γίνεται περισσότερο ώστε πραγματικά να ελοποιηθούν ε, και να δοθεί αυτή η βοήθεια στην Ελλάδα. Ευχαριστώ. Thank you. Thank you, Mrs. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κρέλ. Δεν βλέπω κάποιον εκπρόσωπο από το ECR να θέλει το λόγο. Α, παρακαλώ, παρακαλώ, δεν σας είδα, έχετε το λόγο. Ο κύριος Μαριάς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν είμαι μέλος της Επιτροπής σας αλλά θα ήθελα να θέσω ορισμένα ζητήματα. Καταρχάς, να καλωσορίσουμε και εμείς την κυρία Επίτροπο στην συνεδρίασή μας και να πω το εξής. Πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να προβληματιστεί η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση για το μνημόνιο το οποίο έχει επιβάλει στην Ελλάδα διότι ενώ έχουν δοθεί 240 δισεκατομμύρια ευρώ ως δάνεια τα τελευταία πέντε χρόνια η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει 1,5 εκατομμύριο ανέργους και 40% του πληθυσμού ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας. Άρα λοιπόν το πρόγραμμα απέτυχε και θα αποτύχει και το καινούργιο. Διότι από αυτά τα 86 δισεκατομμύρια το μεγαλύτερο μέρος πηγαίνει για να πληρωθούν τα ομόλογα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα οποία τα αγόρασε με έκπτωση 40%, τα πληρώνεται εις ολόκληρο όλη την ονομαστική αξία και ένα εξοφληθεί και το ΔΝΤ. Άρα από αυτά τα 80 δις στην ελληνική οικονομία, όπως υπολογίζω, ελάχιστα ποσά θα πέσουν, όπως έγινε και από το προηγούμενο. Άρα λοιπόν αυτό να το λάβει υπόψη το Κοινοβούλιο, διότι αυτό το πρόγραμμα, πέραν του ότι είναι αντιλαϊκό, είναι πρόγραμμα λιτότητας, είναι πρόγραμμα μείωσης μισθών και συντάξεων, δεν πρόκειται να βοηθήσει την ελληνική οικονομία, διότι διασώζει απλά τον κύριο Ντράγκη και του πληρώνει όλα τα ομόλογα, τα οποία αυτός πλήρωσε στο 60%. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση. Η περίφημη συμφωνία του Τρίτου Μνημονίου παρανόμως με απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συνέδεσε την εφαρμογή του ΕΣΠΑ και όλων των προγραμμάτων των κοινοτικών με την εφαρμογή του Μνημονίου. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά όλα τα κράτη μέλη έχουν δικαίωμα από τα διαρθρωτικά ταμεία να πάρουν κάποια χρήματα. πουθενά σε κανένα κράτος πλην της ελλάδας δεν συνδέεται αυτό με την εφαρμογή ενός μνημονιακού προγράμματος. άρα είναι μια δεύτερη παραβίαση και αυτό επίσης είναι λάθος. και πάμε τώρα στο τρίτο θέμα είναι πράγματι σωστό και το έχω πει σε πολλές συνεδριάσεις και αυτό πρέπει να εφαρμοστεί όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και ορισμένες χώρες άλλες που είναι σε μνημόνιο ότι πρέπει να αλλάξει η διαδικασία της συγχρηματοδότησης. Διότι όταν με τα προγράμματα τα μνημονιακά στην Ελλάδα αλλά και στα άλλα κράτη επιβάλλεται η μείωση των ελλημάτων η μείωση των ελλημάτων γίνεται κυρίως και το ξέρετε όλοι με τη μείωση των δημοσίων επενδύσεων άρα με τη μείωση των ποσών που διαθέτει ένα κράτος από εθνικούς πόρους για επενδύσεις άρα αδυνατούν τα κράτη αυτά και κυρίως η Ελλάδα να συγχρηματοδοτήσει τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Επομένως δίνονται χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό τον όρο συγχρηματοδότησης. Αυτά τα ποσά δεν υπάρχουν διότι η ίδια η Τρόικα έχει επιβάλει περιορισμούς στην επενδυτική πολιτική και άρα είναι δώρο-άδωρο. Επομένως θα έλεγα στην Επιτροπή και στην προηγούμενη επιτροπή ότι άργησε ότι τέτοιες παρεμβάσεις και τελειώνω I'm going to finish Madam President, τέτοιες παρεμβάσεις σε σχέση με τη συγχρηματοδότηση έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και πολύ καιρό. Όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για τις άλλες χώρες. Άρα εδώ έρχεται πλέον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στηρίξει μια πρωτοβουλία αναγκαία αν θέλουμε να μπορέσουν να εφαρμοστούν τα κοινοτικά προγράμματα. Αυτές είναι οι γενικές παρατηρήσεις που θα ήθελα να κάνω από την πλευρά μου. Ευχαριστώ. Thank you. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ ο κύριος Γιάκοφσιτς, εκ μέρους του Άλντα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα στην Επιτροπή μας. Πάντοτε χαιρόμαστε να μας δίνετε η ευκαιρία να ανταλλάσσουμε απόψεις μαζί σας. Είναι πολύ σημαντική αυτή η στιγμή και είναι κέρια σημασία η παρουσία σας εδώ. για να ανταλλάσσουμε απόψεις και επιχειρήματα και να καταλήξουμε σε αποφάσεις που θα ευνοήσουν την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό. Η πολιτική ομάδα του ΑΛΤΕ είναι υπέρ της άποψης του να χρησιμοποιηθεί η απλουστευμένη διαδικασία χωρίς τροπολογίες και να προσπαθήσουμε να τηρήσουμε όλες τις προθεσμίες, δείχνοντας κατά αυτόν τον τρόπο ότι εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε την προσπάθεια αυτή που απαιτείται για να δοθεί μια νέα ευκαιρία στην ελληνική ανάπτυξη. Τα κονδύλια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την Ελλάδα από τα ταμεία αυτά είναι κονδύλια που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για συγκεκριμένα έργα. και αυτό θα αποτελέσει προϋπόθεση για την έναρξη μιας νέας ανάπτυξης. Τα κονδύλια αυτά δεν θα χρησιμοποιηθούν, όπως είπε ο αγαπητός συνάδελφος από τις τράπεζες, δεν θα τα δώσουμε στον Τράγκη, θα τα χρησιμοποιήσουμε για συγκεκριμένα έργα και ακριβώς αυτό μας ενδιαφέρει και γι' αυτό και το υποστηρίζουμε. Τα 26 δισεκατομμύρια, λέει ο κύριο Μαριάς, θα χρησιμοποιηθούν για τη διάσωση των τραπεζών και για τον κύριο Ντράγκη. Αυτό είπα. Ζητώ συγγνώμη, κύριε Μαριά. Δεν κάνουμε συζήτηση μεταξύ μελών της Επιτροπής. Κύριε Γιάκοψη, συνεχίστε. Ο αγαπητός συνάδελφος δεν κατανόησε πλήρως αυτό που έλεγα. Θα το συζητήσουμε όμως ε, φιλικά πίνοντας τον καφέ μας αργότερα. Ήθελα να πω ότι η παρούσα στιγμή είναι η σωστή στιγμή τώρα που το Κοινοβούλιο καλείται να λάβει μια απόφαση και πρέπει να δείξουμε την αλληλεγγύη μας και τη διάθεσή μας να βοηθήσουμε. δεν λέω ότι μας ικανοποιεί πλήρως η κατάσταση αυτή στην ομάδα των φιλελευθέρων, αλλά στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση που μπορούμε να λάβουμε μια συγκεκριμένη απόφαση, υποστηρίζουμε την προσέγγιση αυτή και θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την απλουστευμένη διαδικασία χωρίς τροπολογίες. Και φαντάζομαι και όλες οι άλλες ομάδες αλληλεγγύη πρέπει να δείξουν προς την Ελλάδα και να κάνουν το ίδιο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σομαζή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε, που ήρθατε στην Επιτροπή μας. Και θέλω κι εγώ να τονίσω ε, την ταχεία αντίδραση της Επιτροπής ε, μετά την διάσκεψη κορυφής. Τώρα πλέον τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα, το, Ευρωπαϊκό, το, Συμβούλιο των Υπουργών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει επίσης ε, να δείξουν την ίδια ε, ταχεία αντίδραση και να κατανοήσουν τον επίγοντα χαρακτήρα. Διότι αντιμετωπίζουμε μία κατάσταση έκτακτης ανάγκης και πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας και στη δική μας Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Υπάρχει επίγον χαρακτήρας διότι εάν η Ελλάδα δεν εφαρμόσει πάρα πολύ γρήγορα ορισμένα επιχειρησιακά προγράμματα ε, για την περίοδο 2007-2013 μιλάμε για 2 δισεκατομμύρια πιστώσεων τα οποία θα χαθούν. Και γνωρίζουμε όλοι ότι η Ελλάδα χρειάζεται επιγόντως ρευστότητα. Όλοι γνωρίζετε πως έχει η κατάσταση. Νομίζετε ότι θα ήταν προς τιμήν των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και δεν θα ήταν περίεργο το να χαθούν τα 2 δισεκατομμύρια αυτά για την Ελλάδα υπό τις παρούσες προϋποθέσεις. Εμείς πρέπει να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες για να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Εφόσον έχουμε επίγουσα κατάσταση ή εξαιρετική κατάσταση, θα πρέπει να ληφθούν και εξαιρετικά και επίγοντα μέτρα. Και γι' αυτό η δική μας πολιτική ομάδα είναι υπέρ της απλουστευμένης διαδικασίας χωρίς τροπολογία. Μέτρα έκτακτης ανάγκης λοιπόν και επί της ουσίας, ακριβώς ε, όπως η πρόταση κανονισμού της Επιτροπής. Όπως και εσείς κύριε Επίτροπε, επιμένω κι εγώ ότι αυτή η πρόταση είναι δημοσιονομικά ουδέτερη, δηλαδή δεν κοστίζει περισσότερα χρήματα στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης η πρόταση αυτή. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σαφής η θέση της δικής μας πολιτικής ομάδας, της Ενωτικής Αριστεράς. Δηλαδή θέλουμε να εφαρμοστεί το άρθρο 51 του κανονισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Βάνα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε, κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα και εγώ να σας καλωσορίσω στην Επιτροπή μας. Και εμείς οι πράσινοι χαιρετίζουμε ε, το πακέτο αυτό το οποίο μας προτείνεται ως έκτακτο πακέτο μέτρων. Ξέρουμε ότι δεν θα λύσει τα προβλήματα της κρίσης στην Ελλάδα αυτό το πακέτο μέτρων, αλλά είναι απόλυτα απαραίτητο για τις επενδύσεις και συγκεκριμένα τα διαρθρωτικά ταμεία μας έχουν δείξει τα τελευταία χρόνια ότι ότι ε, δεν υπήρχαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις ε, συμμετοχής και της ελληνικής πλευράς. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη της ε, ελληνικής οικονομίας και για την τεχνική βοήθεια η οποία προτείνεται. Είναι αυτά τα κονδύλια απαραίτητα για την υλοποίηση των προγραμμάτων στην Ελλάδα. Συνολικά είναι λίγα τα χρήματα, δεν είναι επιπλέον χρήματα τα οποία δίδονται. Εμείς όμως εδώ προσπαθούμε να συνεννοηθούμε για αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα και αυτή τη στιγμή έχουμε μια επίγουσα κατάσταση, επίγοντα μέτρα και πρέπει να δράσουμε γρήγορα και να χρησιμοποιήσουμε μια ε, επίγουσα διαδικασία. Εμείς ως ε, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουμε ευθύνη και πρέπει να δράσουμε γρήγορα. Σας ευχαριστώ και για την ταχεία υποβολή της πρότασης της Επιτροπής και βεβαίως και εμείς προτιμούμε την απλουστευμένη διαδικασία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Νταμάτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την Επίτροπο για την παρουσία τη. Μας ενημέρωσε για την τροποποίηση του κανονισμού Βλέποντας την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα δεν μπορούμε να μην δεχθούμε θετικά το αίτημα για προχρηματοδότηση 2007-2013 ή μάλλον για την περίοδο 2014-2020. Πάντα η ομάδα μας υποστήριξε να υπάρξει μια μεγαλύτερη ευελιξία απέναντι στον ελληνικό λαό ασκώντας κριτική στις πολιτικές λιτότητας και στους όρους που έχουν επιβληθεί στην Ελλάδα. Πραγματικά θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να βγάλουμε εντελώς και να μην συνυπολογίζεται η συγχρηματοδότηση στο έλλειμμα. Νομίζω λοιπόν ότι στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής θα πρέπει να δούμε ότι η Ελλάδα έχει ένα καλό επίπεδο απορρόφησης, ποσοστό απορρόφησης των διαφορετικών ταμείων και θα μπορέσουμε έτσι να καθησυχάσουμε και τις χώρες μέλη που έχουν κάποιες δίσταγμους διότι δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση κάποια δημοσιονομική αλλαγή. Δεν υπάρχει κάτι, είναι ουδέτερο εντελώς για τις πληρωμές οι οποίες προβλέπονται στα πλαίσια του πολιετούς πλαισίου. Η συγχρηματοδότηση λοιπόν για το διαφθρωτικό ταμείο, για το κοινωνικό ταμείο και για το ταμείο συνοχής θα παραμείνει ως έχει. Είμαστε υπέρ λοιπόν της απλουστευμένης διαδικασίας χωρίς τροπολογίες. Ευχαριστούμε κύριε Ανταμάτο. Κύριε Μπουνάν, θα θέλετε να ε, πάρετε το λόγο εκ μέρους της ομάδας σας. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Για μα είναι προφανές ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, φέρεται σαν πυρομανής πυροσβέστης με την Ελλάδα διότι η κρίση η οποία πλήττει την Ελλάδα είναι απόρρια των πολιτικών λιτότητας που της έχει επιβάλει η Επιτροπή μεταξύ άλλων και οι ε, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκηση αυτή τη στιγμή δεν έχουν καν τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν το 5% των επενδύσεων ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, Πυρομανή πυροσβέστη λοιπόν και ο κ. Γιούγκερ που προσπαθεί να σβήσει μία φωτιά την οποία δεν, της οποίας δεν έχει πλέον τον έλεγχο. Εν ολίγης, η Ευρωπαϊκή Ένωση με το ένα χέρι δίνει αυτά τα οποία παίρνει με το άλλο χέρι. Αυτό το οποίο λοιπόν προτείνουμε για την Ελλάδα δεν θα έχει τα προτινόμενα αποτελέσματα. Ε, η Ελλάδα είναι μια χώρα που ε, βρίσκεται στην ασφυξία του χρέους της ε, μέσα στο κοινό νόμισμα το ευρώ. Επομένως, γιατί να χρησιμοποιήσουμε ευρωπαϊκά κονδύλια για να χρηματοδοτήσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο δεν θα σταματήσει την ελληνική αιμορραγία και δεν ε, θα εφαρμόσει τα, τελικά τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Ακούσαμε ε, στην Επιτροπή μας τα διάφορα επιχειρήματα. Ε, έχουμε ακούσει και τα επιχειρήματα για την αναδιάθρωση του χρέους Έχουμε ε, καθυστερούμενες πληρωμές πάνω από 20 δισεκατομμύρια για το 2015. Τι θα επιτύχουμε με το 1 δισεκατομμύριο το οποίο ε, απελευθερώνουμε για την Ελλάδα. Πιστεύω ότι ανοίγουμε το κουτί της πανδώρας με ένα τέτοιο μέτρο, διότι πολλά κράτη θα αρχίσουν να ζητούν κατεξαίρεση ενισχύσεις με συγχρηματοδότηση Νομίζω λοιπόν ότι οι απαντήσεις που προσπαθείτε να δώσετε δεν είναι στο ύψος των προβλημάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίσουμε, συνεχίζουμε τώρα με τα μέλη της Επιτροπής Ρέτζη που έχουν ζητήσει το λόγο. Στον κατάλογο των μιλητών έχω καταρχήν την κυρία Σπυράκη. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους. Σήμερα η Επιτροπή προτείνει μια εξαιρετική διάταξη για τη χώρα μας που θα επιτρέψει στην Ελλάδα να πάρει μια βαθιά ανάσα και να συνεχίσει στο δύσκολο δρόμο που έχει μπροστά της. Η παρέμβαση αυτή την οποία προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εάν συνοδεύεται από ένα απλουστευμένο πλαίσιο και από κατάλληλη θεσμική ενίσχυση, θα μπορούσε να δώσει μια όθηση ρευστότητας και με άμεσες ε, ε, συνεισφορές Υπότιτλοι Authorwave για να καλυφθεί το κενό που υπάρχει μεταξύ του προηγουμένου και του τωρινού πολιετού ε, προγράμματο. Ξέρετε αγαπητοί συνάδελφοι ότι στι 20 Σεπτεμβρίου έχουμε εκλογέ στην Ελλάδα και σύμφωνα με τι τελευταίε δημοσκοπήσεις τα δύο πρώτα κόμματα, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, είναι ε, πολύ κοντά το ένα με το άλλο. Θα ήθελα να μιλήσω εκ μέρου τη δική μου πολιτική ομάδα, εκ μέρους του κόμματο τη Νέα Δημοκρατία. Ε, χρειαζόμαστε αυτέ τι διαφορετικές μεταρρυθμίσεις και πρέπει να μα δοθεί ο τρόπος να ρυθμίσουμε τα προβλήματα της οικονομίας χωρίς να καθυστερούμε καθόλου. Καταλαβαίνω ότι και άλλα κράτη-μέλη έχουν επίγουσες ανάγκες, αλλά σήμερα είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της Ελλάδας. Και δεν συμφωνώ να ακολουθήσουμε την απλουστευμένη διαδικασία και να δώσουμε στην Ελλάδα μια ευκαιρία το ταχύτερο δυνατόν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ξέχασα να αναφέρω ότι τώρα που λαμβάνουν το λόγο τα μέλη της Επιτροπής το όριο είναι δύο λεπτά. Κύριε Σπυράκη, σας ευχαριστώ γιατί τήρησατε το χρόνο σας. Κύριε Μπρέσσε. Ε, Δεν θα ήθελα να πω κάτι για τη διαδικασία γιατί η συντονίστρια μας ήδη εξέφρασε την ομάδα και συμμερίζομαι απολύτως την άποψή της. Θα ήθελα όμως το λόγο για το εξής. Πάρα πολύ συχνά οφείλουμε να τροπολογήσουμε ουσιαστικά να αλλάξουμε τις συγχρηματοδοτήσεις στην περιφερειακή πολιτική όταν υπάρχει κάποια κρίση. Θα πρέπει η Επίτροπος λοιπόν να μας πει αν δεν θα πρέπει να περάσουμε σε μια πιο διαφορετική αλλαγή που να επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν υπάρχουν ε, εγγυήσει ε, για μειωμένες έστω εγγυήσει να μπορεί να το κάνει αυτό χωρίς να τροποποιούνται οι κανόνες συνεχώς. Γνωρίζουμε ότι η συγχρηματοδότηση των τοπικών αρχών και των κρατών όταν υπάρχει μια κάποια κρίση αντιμετωπίζει δυσκολίες. Όλοι γνωρίζουμε επίσης ότι σε εποχές κρίσης ε, μειώνονται οι επενδύσεις και δεν θα πρέπει να μειώνονται οι τρέχουσες δαπάνες. Πρέπει λοιπόν να τροποποιηθούν οι κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, τροποποιώντας ε, την αντιμετώπιση των επενδύσεων αντίστοιχα με τις τρέχουσες. Γνωρίζω ότι θα πρέπει να αφαιρεθούν επίσης οι επενδύσεις από τον υπολογισμό των ελλημάτων και για μια ακόμη φορά στην ουσία εδώ αποδεικνύεται ότι αν δεν τροποποιηθούν σε διαρθρωτικό επίπεδο τα θέματα που άπτονται του κοινοτικού προϋπολογισμού τότε σαν συνέπεια έχουμε τον κίνδυνο για τις χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες να βλέπουν τις επενδύσεις τους να συντρίβονται και αυτό δεν βοηθάει στην ανάκαμψη της οικονομίας. Ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ ε, ε, πρόεδρε ε, και κυρία Επίτροπε. Ε, ε, αντιλαμβάνομαι ακριβώ το τι περνάει ο ελληνικό λαό αυτή την περίοδο, γιατί σα διαβεβαιώ ότι και στη Βουλγαρία τα πράγματα δεν είναι πολύ καλύτερα. Ε, είμαι σίγουρο ότι η Ελλάδα χρειάζεται τη βοήθειά μα και πάντοτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο διαφύλαται την αρχή τη αλληλεγγύη ε, πάντοτε δηλαδή ήταν υπέρ του να υποστηρίζει το ταχύτερο δυνατό και η απόδειξη είναι και τα σχετικά ταμεία που υπάρχουν όπως το Ταμείο Συνεχής και ούτω καθεξής ε, και, ε, και το Κοινοβούλιο λοιπόν έχοντας παίξει πάντοτε ένα τόσο ενεργό ρόλο σε αυτές τις διαδικασίες θα πρέπει να το κάνει και για μία ακόμα φορά τώρα. Ε, θεωρώ όμως ότι θα πρέπει να εμείνουμε στην άποψή μας και κατά συνέπεια θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να θέσουμε ερωτήματα στην Επιτροπή στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας. Ναι, να κινηθούμε όσο γίνεται ταχύτερα στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, αλλά ε, εμείς για παράδειγμα ήμασταν η πρώτη κοινοβουλευτική επιτροπή η οποία είχε ψηφίσει υπέρ των ε, διαφθορτικών και επιδοτικών ε, ταμείων. Οπότε καλό θα ήταν να έχουμε και σε αυτό το πλαίσιο αυτής της διαδικασίας τη δυνατότητα να θέσουμε ερωτήματα για να αλλάξουμε και ό,τι χρειάζεται να τροποποιηθεί. Ε, εγώ ήμουν υπέρ διαφόρων αλλαγών οι οποίες δεν αφορούσαν καν τη Βουλγαρία για πολλές χώρες. Ε. Για παράδειγμα παρεκκλήσεις από το 1 1, 1 3 και ε, ούτω καθεξής. Αλλά νομίζω πως τώρα εδώ θα πρέπει να εστιάσουμε λίγο όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε κάποια άλλα κράτη-μέλη στο ποιες απαντήσεις ε, μπορούμε ε, να δώσουμε. Δηλαδή το τι σκέφτονται τα κράτη-μέλη μας ε, και σήμερα αλλά και τι αύριο, αν για παράδειγμα ακολουθήσει κάποιο άλλο κράτος μέλος, χρειαστεί κάτι αντίστοιχο. Άρα λοιπόν είμαι υπέρ του να υποστηρίξουμε την Ελλάδα το ταχύτερο δυνατό και όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και άλλα κράτη-μέλη τα οποία πλήττονται από τις συνέπειες της κρίσης. Ευχαριστώ. Δύο παρατηρήσεις για να προσθέσω και εγώ στη συζήτηση. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε γρήγορα. Η διαδικασία χωρίς τροπολογίες είναι η σωστή. Ταυτόχρονα θα ήθελα να πω στους φίλους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ότι θα πρέπει εμείς να ανακτήσουμε ένα πιο δραστήριο ρόλο του Κοινοβουλίου, όχι για την Ελλάδα ειδικά, αλλά για τέτοιου είδους περιπτώσεις και θέματα. Είναι κάτι το οποίο έτσι κι αλλιώς ε, καλούμεθα να συζητήσουμε τους επόμενους μήνες. Το θέμα δηλαδή το πώς θα ξεπεράσουμε το μηχανισμό της Τρόικα με έναν πιο δραστήριο ρόλο του Κοινοβουλίου ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα πρέπει να είναι πιο αποφασιστικός. Το να βιαστούμε τώρα δεν σημαίνει ότι δεν θα συζητήσουμε τα προβλήματα τα οποία έχουμε. Σημαίνει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μην παγώσουν οι διαδικασίες οι οποίες έχουν ξεκινήσει. Εμείς θέλουμε να διεκδικήσουμε έναν σοβαρότερο ρόλο του Κοινοβουλίου να είμαστε το εμπόδιο στην διαδικασία της εφαρμογής του μηνός Ιουλίου. Πρέπει λοιπόν να βιαστούμε, πρέπει να δεχθούμε την πρόταση της Επιτρόπου και της Επιτροπής και ταυτόχρονα να μην χάσουμε θα έλεγα τα θέματα τα οποία έχουμε κληρονομήσει γύρω από τους τομείς αυτούς. Ρωτώ λοιπόν την Πρόεδρο και την Επίτροπο Μπορούμε να δημιουργήσουμε ίσως ένα δικό μας μνημόνιο γύρω από τα θέματα αυτά. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι ιταλικό, είναι και σε άλλες χώρες. Η προσθετικότητα δεν ισχύει για πάρα πολλές χώρες η προσθετικότητα. Πρέπει να το συζητήσουμε, όχι μόνο για την Ελλάδα. Είναι ένα ευρωπαϊκό θέμα. Το θέμα του διαχωρισμού ανάμεσα στις, επενδυτικές, ε, στις επενδύσεις ε, και τις πιστώσεις αποκλειστικά για επενδύσεις και τις ε, πιστώσεις για την κάλυψη των τρέχουσών δαπανών πρέπει να το ξεχωρίσουμε αυτά τα δύο, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν από τη συζήτηση αυτή να μην ε, κάνουμε μια αντιπαράθεση η οποία θα καθυστερήσει. Πρέπει όμως αντίθετα να θέσουμε το Κοινοβούλιο σε θέση να αναλάβει τις ευθύνες του, να λαμβάνει αποφάσεις ταχύτητα και να μην απολέσουμε τα θέματα αυτά τα οποία πρέπει να συζητήσουμε. Πρέπει λοιπόν σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να συζητήσουμε το μέλλον αυτών των θεμάτων γιατί θα τα δούμε μπροστά μας τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια. Αν καθυστερήσουμε τις συζητήσεις το λάθος θα είναι διπλό. Μπορούμε λοιπόν πρώτον να αποφασίσουμε σήμερα να προχωρήσουμε γρήγορα και ταυτόχρονα να συνεχίσουμε με μεγάλη ταχύτητα τις συζητήσεις με την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ. Μπάγκοβιτς. τα, τα δικαιώματα της ελεύθερης κυκλοφορίας και ε, το κοινό νόμισμα θα ήθελα να πω ότι είναι δύο από τις ε, βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Και, αντιλαμβανόμαστε ότι τα μία ταμεία είναι κέρια σημασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για επενδύσεις σε κράτη-μέλη τα οποία έχουν υποστεί της επιπτώσης μιας κρίσης. Η Ελλάδα αποτελεί βέβαια ένα παράδειγμα Ενό ε, τέτοιου κράτους Οπότε ε, για την περίοδο 2015-2016 θα πρέπει να αυξήσουμε την βοήθειά μας ε, προ την Ελλάδα. Η πρόταση λοιπόν για μια απλουστευμένη διαδικασία και επιταχυμένη διαδικασία ούτω ώστε να ρεύσουν το ταχύτερο δυνατό τα επενδυτικά κονδύλια στην Ελλάδα είναι η σωστή απόφαση και μπορώ να την υποστηρίξω. Έχουμε συζητήσει στο παρελθόν την οικονομική κρίση στην Ελλάδα, έχουμε συζητήσει και την κρίση του ευρώ, ειδικότερα σε σχέση με την Ελλάδα, αλλά αυτή τη στιγμή η Ελλάδα αντιμετωπίζει και, και μια κρίση σε ό,τι αφορά τους πρόσφυγες, οπότε σίγουρα θα πρέπει να την ε, βοηθήσουμε το ταχύτερο δυνατό. Ε, ο κύριος Βαν Μίλτερ που έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, θα μιλήσω στο γλωσσό του κ. Βανίστερο, ούτε ώστε να μην υπάρξουν παρανοήσει. Να πω ε, λοιπόν πω με λίγο με την ε, θέση του Λαϊκού Κόμματο. Ε, δηλαδή, ε, έχουμε μια απλουστευμένη διαδικασία την οποία θέλουμε να ακολουθήσουμε τελικά ποιο είναι, ποια είναι η αντίρρηση που θα μπορούσατε να έχετε, να έχετε στην πρόταση αυτή της Επιτροπής ώστε να υποβάλλετε από τη δική σα πλευρά τροπολογίας. Μας είπατε δηλαδή ότι θέλετε μια ε, κανονική διαδικασία, τόσο ώστε να έχετε δυνατότητα να υποβάλλετε τροπολογίε. Οπότε θέλουμε να ακούσουμε και το υπόλοιπο του, του χρόνου μα σα το δίνω για να απαντήσετε στον κύριο Βανίστερο. Okay. Ε, I, like to, not to answer now, nu niet geen antwoord te geven, maar dat in de... Δεν θα απαντήσω τώρα, σε αυτό με ρωτήσατε, αλλά στο τελικό γύρο των παρεμβάσεών μας, όπου θα πρέπει να λέμε και μια απόφαση, θα σας απαντήσω σε αυτό που με ρωτήσατε. Πρόεδρος εκτός μικροφώνου. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ελλάδα επλήγει ε, πάρα πολύ από την πολιτική λιτότητα και από την ε, Τρόικα και μάλιστα η σημερινή Επιτροπή και το σημερινό Κοινοβούλιο θεωρούν όπως αποτέλεσαν ε, σφάλματα τα όσα αποφασίστηκαν. Επίσης η Ελλάδα υπήρξε το θύμα ε, δύο κλεπτοκρατικών ε, δυναστεών ε, και μετά ήρθε και η Τρόικα με αποτέλεσμα να οδηγηθεί σε μια εξαιρετική κατάσταση για την οποία χρειαζόμαστε και εξαιρετικά μέτρα οπότε θα πρέπει να αποδεχθούμε την απλουστεμένη ταχύτερη διαδικασία όπως αυτή προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ας διερευνήσουμε και τις υπεραιτέρω δυνατότητες που έχουμε σύγχρηματοδότησης οι οποίες βέβαια μπορούν να αφορούν και άλλα κράτη-μέλη, όχι μόνο την Ελλάδα, σε ένα μεταγενέστερο στάδιο. Ένα κάπω ανόητο ερώτημα θα ήθελα να θέσω. Δεν μπορώ να αντιληφθώ αυτό που συμβαίνει σήμερα. Δηλαδή, η Ελευθερία Νασιονάλ και το ΕΛΚ είναι κατά της ε, διαδικασία, διαδικασίας, της διαδικασία, επειδή έχουμε ε, τις ε, πρόορες εκλογές ε, στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ποια είναι δηλαδή το πολιτικό μήνυμα το οποίο δίνουν για παράδειγμα αυτές οι πολιτικές ομάδες στους Έλληνες πριν από αυτές τις εκλογές οι οποίες έρχονται σύντομα στην Ελλάδα. Οπότε ως Ρουμάνος και ως σοσιαλιστής σε κάθε περίπτωση είμαι 100% υπέρ της πρόταση της Επιτροπής για ταχύτερη διαδικασία. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριος Μασκό. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν θα μιλήσω επί της διαδικασίας, διότι συμφωνώ απολύτως με την συντονίστρια που έλαβε το λόγο εκ μέρους της πολιτικής μας ομάδας. Συμφωνώ, και αυτό θέλω να πω, ότι συμφωνώ να δράσουμε κατεπήγοντος. Πρέπει να βοηθήσουμε την Ελλάδα να σωθεί, πρέπει να δημιουργήσουμε γρήγορα ειδικού μηχανισμούς για την Ελλάδα η ερώτηση που θέλω να κάνω είναι η εξή: Πριν από λίγα χρόνια ξαναδώσαμε δισεκατομμύρια στην Ελλάδα και εμείς ως πολιτικοί υπεύθυνοι, ως ερετοί ε, έχουμε το καθήκον να πούμε τι πρέπει να γίνει ούτω ώστε αυτά τα χρήματα που είναι πολύ σημαντικά, αυτά τα χρήματα που θα δοθούν πώς θα γίνει να φτάσουν στα σωστά χέρια δηλαδή αυτοί οι οποίοι υποφέρουν, αυτοί οι οποίοι έχουν δυσκολίες να υποφεληθούν από τα χρήματα αυτά αυτή είναι η ανησυχία μας, διότι μπορεί να έχουμε εμπιστοσύνη σε οποιαδήποτε κυβέρνηση κερδίσει τις εκλογές, αλλά θα πρέπει να, να υπάρξει κάτι, μια έκθεση αξιολόγησης, μια ενδιάμεση έκθεση, για να μπορέσουμε να αξιολογούμε εμείς κάθε χρόνο την κατάσταση, για να μην χρειάζεται τρία χρόνια αργότερα να επανέλθουμε στα ίδια προβλήματα που γνωρίζαμε στο παρελθόν. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ρένκε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κυρία Επίτροπε, που ήρθατε στην Επιτροπή μας. Δεν θέλω κι εγώ να μπω στα διαδικαστικά της υπόθεσης. Πιστεύω ότι αν δεν ακολουθήσουμε την ταχεία διαδικασία δεν θα υπάρχει πλέον το θετικό μήνυμα από την ταχεία υποβολή της πρότασης της Επιτροπής. Το ερώτημα δεν είναι μόνο του αν θα γίνουν οι επενδύσεις και πότε θα γίνουν οι επενδύσεις. Ε, είναι σημαντικό και το σε τι θα γίνουν επενδύσεις. Ήμουν στην Ελλάδα τέλος Ιουλίου και μίλησα με τις τοπικές αρχές αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα και μου έλεγαν ότι πολύ συχνά δεν έχουν τη δυνατότητα, δεν έχουν τις διοικητικές δυνατότητες εφαρμογής και υλοποίηση των προγραμμάτων των διαθροτικών ταμείων. Εποφελούμε τη παρουσία τη Επιτρόπου στην Επιτροπή μα και θα ήθελα να ρωτήσω για τα, προβλήματα τεχνικής, για τα προγράμματα τεχνική βοήθεια. πώς προτείνει η Επιτροπή να βοηθήσουμε τις αρχές στην Ελλάδα να εφαρμόσουν τα προγράμματα. Γιατί ακόμη και με την ταχεία διαδικασία οι ελληνικές αρχές θα έχουν πολύ μικρό χρόνο στη διάθεσή τους για να απορροφήσουν τα κονδύλια και είναι πάρα πολύ σημαντικό η Επιτροπή να στείλει προσωπικό στην Ελλάδα, να δημιουργήσει δυνατότητες, να δημιουργήσει ικανότητες επιτόπου, ώστε να επενδυθούν τα χρήματα εγκαίρως και να επενδυθούν σε βιώσιμα προγράμματα και πιστεύω ότι δεν είναι μόνο θέμα επένδυσης, είναι θέμα επένδυσης ε, με βιώσιμο τρόπο σε σωστά προγράμματα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε η Επίτροπος να μας δώσει κάποιες λεπτομέρειες για το πώς έχετε προγραμματίσει τεχνική βοήθεια. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μισελ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε και κυρία Επίτροπε. Ήδη ελέγχθησαν πολλά και συμφωνώ με, ε, εν με αυτά που είπε η κυρία Χέιλ. Ε, Νομίζω ότι αυτή τη συζήτηση την οποία διεξάγουμε εδώ δεν θα πρέπει να την ε, διεξάγουμε στο πλαίσιο ιδεολογικής ή προεκλογικής συζήτησης. Μερικές φορές έχουμε την εντύπωση ότι χρησιμοποιούνται αυτά τα θέματα είτε για καθυστέρηση είτε για προεκλογικές συζητήσεις. Αυτό το οποίο ε, ε, θέλω να πω είναι ότι ορισμένοι ομιλητές ε, μιλούν σαν να πρόκειται να στείλουμε κάποιο δωράκι στην Ελλάδα. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω, να υπενθυμίσω σε όλους ότι σε αυτή την αίθουσα πολύ συχνά έχουμε συζητήσει το πώς πρέπει να γίνεται αποτελεσματικά η υλοποίηση των διαθροτικών κονδυλίων. Και όλοι συμφωνούμε ότι χρειάζονται κάποιοι μηχανισμοί και οι φυστάμενοι μηχανισμοί σε πολλές περιπτώσεις πρέπει να τροποποιηθούν για να βρούμε έναν τρόπο ε, που θα είναι πιο εύκολος Ακούτε επιχειρήματα που λένε ότι ε, αν ε, το κάνουμε αυτό για την Ελλάδα ε, θα έρθουν και άλλες χώρες να το ζητάνε. Μα είναι αυτονόητο. Αν είμαστε επιτυχημένοι σε αυτό το οποίο κάνουμε θα έρθουν και άλλες χώρες να ζητούν την εφαρμογή επιτυχημένων μέτρων. Εγώ θέλω να σας παρακαλέσω για άλλη μια φορά να σκεφτείτε ότι εδώ έχουμε ένα θεμελιώδες ερώτημα. Τι κάνουμε με τα κονδύλια ούτως ώστε να είναι αποτελεσματικά και να φτάνουν εκεί όπου πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Και η κυρία Κρέτσου είπε ότι ε, τον Ιούλιο συζητήθηκε αυτό το θέμα, ότι δεν φτάνουν τα κονδύλια στους σωστούς δικαιούχους στην Ελλάδα. Τι κάνει η Επιτροπή γι' αυτό και ε, πώς θα φροντίσουμε εμείς ως ευρωβουλευτές να μην ε, φρενάρουμε τη διαδικασία αλλά να συμβάλλουμε ώστε τελικά όντως να συμβεί αυτό το οποίο επιθυμούμε. Ευχαριστώ πολύ. κυρία Λατίτσου. Ευχαριστώ Πρόεδρε και σας ευχαριστώ Επίτροπε για την παρουσία σήμερα εδώ. Νομίζω πως αυτή η πρόταση από την πλευρά της Επιτροπής είναι ε, και πολύ καλή και απαραίτητη. Δεν θα ε, είναι τώρα την βέβαια τη συζήτηση που κάνουμε σε σχέση με άλλα κράτη-μέλη, γιατί θα πρέπει και εκεί να δούμε πώς θα πρέπει η υλοποίηση να γίνεται καλύτερα, ειδικότερα των πολιτικών συνοχής, επιτόπου σε όλη την Ευρώπη, αφού έχουμε και μία σειρά από κράτη-μέλη ε, που βρίσκονται σε δυσκολίες. Ε, και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι δεν θα πρέπει να αναλαμβάνουμε δράση ε, μόνο όταν μια χώρα βρίσκεται ήδη σε προβλήματα όπως στην περίπτωση της Ελλάδας για να αλλάξουμε κάτι στον κανονισμό. Κάτι δηλαδή, εδώ πρόκειται για κάτι το οποίο θα πρέπει να, να είχαμε συζητήσει και προηγουμένως. Εν πάση περιπτώσει εδώ θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι για την ε, περίοδο 2017-2013 προτείνουμε να αυξήσουμε την προχρηματοδότηση ή μάλλον την συγχρηματοδότηση ε, μέχρι το 100%. Αλλά θα πρέπει εδώ να λάβουμε υπόψη μας ε, ότι πρόκειται για το 100% του επιλέξιμου τμήματος ε, του προγράμματος και το υπόλοιπο λοιπόν του πραγματικού κόστος προγράμματος θα πρέπει η Ελλάδα να, να δει πώς θα το καλύψει. Αλλά από εκεί και μετά ο ρόλος του EIP ή άλλων μηχανισμών έρχεται εδώ να εξεταστεί για το πώς θα καλυφθεί το υπόλοιπο αυτού του επενδυτικού προγράμματος. Θα ήθελα απλώς να το αναφέρω αυτό. Το 100% αφορά το επιλέξιμο τμήμα. Μετά πάλι ε, αυτήν την ε, περίοδο 2007-2013. Δηλαδή έχουμε εκεί τη μία περίοδο και μετά 2014-2015 άλλη διάσταση με αύξηση του ποσοστού προχρηματοδότηση ώστε η Ελλάδα να είναι σε θέση να λάβει περισσότερα κονδύλια ως προχρηματοδότηση. Εδώ λοιπόν πώς ε, τίθεται το ερώτημα, θα βοηθήσουμε στην υλοποίηση αυτών των επενδύσεων. Δηλαδή πώς θα διασφαλίσουμε ε, το ότι η Ελλάδα θα χρησιμοποιήσει πράγματι αυτά τα χρήματα και όχι να έχουμε τελικά μία απορρόφηση και επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση 21η Δεκεμβρίου του 2016 εκμεώτος αυτών των κοντιλίων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα για να συζητηθεί. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος ή Πρόεδρος, συγγνώμη, ο κ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο. Δεν θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση ή αυτά τα οποία είπε έτσι και ο συντονιστής μας. Είναι υποχρεωτικό ε, να προχωρήσουμε στη βοήθεια. Δεν μιλάμε βέβαια για ανθρωπιστική βοήθεια προς τον ελληνικό λαό, αλλά μιλάμε, αυτό θα ήταν υποτιμητικό κατά κάποιο τρόπο. Το θέμα είναι να μιλήσουμε για έκτακτη βοήθεια και το πώς η έκτακτη βοήθεια αυτή θα εγκριθεί από τις διαδικασίες των κοινωτικών οργάνων. Συμφωνώ με την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πλήρως λοιπόν. Θα ήθελα να τονίσω εδώ αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα τα οποία είπε ο συνάδελφος Μόσκου και ε, η Γερμανίδα συνάδελφος. Αφού συμφωνήσω μαζί τους θα ήθελα να πω ότι και σε επίπεδο τεχνικό και σε επίπεδο πολιτικό αυτό το οποίο έχει σημασία αυτή τη φορά η διαδικασία αυτή να λειτουργήσει έχει μεγάλη σημασία να ικανοποιήσει τις ανάγκες που έχει ο ελληνικός λαός και ε, η, ίδια η ελληνική δημοκρατία και οι θεσμοί της ελληνικής δημοκρατίας. Είναι απαραίτητο στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν να υπάρξει ένα σύστημα ελέγχου αναμεμειγμένο με τη βοήθεια έτσι ώστε τα χρήματα αυτά να μην χρησιμοποιηθούν σωστά, να μην ξοδευτούν και στην ουσία να μην χρησιμοποιηθούν. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να τα όλα αυτά, δεν ξέρω μέσω μιας επιτροπής ειδική, μέσω εξαμήνων εκθέσεων, να υπάρχει όμως έλεγχος έτσι ώστε οι πιστώσεις αυτές να πάνε εκεί που χρειάζεται, στον ελληνικό λαό. Το πρόβλημα αυτό δεν είναι μόνο ένα πρόβλημα αυστηρά ελληνικό. Αν χρειάζεται αυτό το σύστημα θα πρέπει να μπορούμε να είμαστε σε θέση σε επίπεδο διοικητικό θεσμικό να χρησιμοποιούμε τα μέσα τα οποία χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν. Νομίζω ότι η ορολογία την οποία χρησιμοποιούμε είναι ότι όλα αυτά μπορεί να συμβούν και σε άλλες χώρες. Αυτό είναι κανόνας του παιχνιδιού. Πρέπει να μπορούμε να βοηθήσουμε λοιπόν και θα πρέπει έτσι ώστε ε, να βελτιώσουμε την ίδια τη λειτουργία των θεσμών μας για να βοηθάμε αποτελεσματικότερα. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Τελευταίος ομιλητής, Ροντρίγκες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως ξέρετε προερχόμαι από την Πορτογαλία. Πρόκειται για μια χώρα η οποία σφαγιάστηκε από τη λιτότητα. Με κορύφωση αυτής της διαδικασίας τη μεγάλη φτώχεια που επικρατεί στη χώρα μου πλέον. Έχουμε πάρα πολλές αμφιβολίες εμείς οι Πορτογάλοι για την χρησιμότητα αυτού του είδους των επιδοτήσεων, των επενδύσεων μάλλον. Μια τεχνική βοήθεια είναι πάρα πολύ σημαντική βέβαια στον τομέα αυτό όταν επικρατεί λιτότητα. Από την άλλη όμως θα πρέπει να προσέξουμε έτσι ώστε να υπάρχει ένα απλοποιημένο καθεστώς που θα διέπει τις επενδύσεις. Λοιπόν αυτά δεν νομίζω ότι θα ήθελε κάποιος άλλος το λόγο. Α, ο κύριος Βανίστελ Ρόι θέλει να δώσει μια απάντηση. Ναι, θα ήθελα να, να ρωτήσω πώς, τι μέθοδο θα ακολουθήσουμε για να πάρουμε την απόφαση. Πρώτα θα πρέπει να ακούσουμε την Επίτροπο, έτσι δεν είναι. Καλώς τώρα με την κατάληξη της συζήτησης αυτής επιτρέψτε μου και εμένα να κάνω κάποια σχόλια σαν πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης. Είναι σημαντική η συνάντηση αυτή, αν και είναι έκτακτη όπως είπαμε, είναι σημαντική γιατί προσπαθούμε να λειτουργήσουμε με ευθύνη, προσπαθούμε να αναλάβουμε την ευθύνη των καθηκόντων μας και να λύσουμε τα προβλήματα στην Ευρώπη με τον δυνατό και καλό τρόπο, κατάλληλο τρόπο σαν κοινοβούλιο. Θα ακολουθήσουμε και θα στηρίξουμε την απλοποιημένη διαδικασία δεν είμαστε υπέρ μιας διαδικασίας η οποία θα είναι αδιαφανής και ανεξέλεγκτη χωρίς δυνατότητες τροπολόγησης. Όχι, αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να είμαστε κυρίως αποτελεσματικοί. Σε άλλες περιπτώσεις, και αυτή είναι προσωπική μου γνώμη, ε, αν δεν το κάνουμε αυτό δηλαδή, τότε ο χρόνος που θα χαθεί θα είναι πάρα και στις συζητήσεις τις κοινοβουλευτικές που έχουμε ε, δεν θα υπάρξει αποτέλεσμα και δεν θα υπάρξει και πολιτική δήλωση για τη στήριξη ουσιαστικά της Ελλάδας. Αλλά θα συμφωνήσω και με όλους τους συναδέλφους οι οποίοι ε, υπογράμμισαν τον ρόλο του Κοινοβουλίου στον έλεγχο της διαδικασίας και στο ότι θα πρέπει να μάθουμε ε, το τι συνέβη σε κάθε χώρα και να το χρησιμοποιήσουμε. Πιστεύω ότι από κοινού θα μπορέσουμε να ελέγξουμε την κατάσταση στην Ελλάδα και έτσι να παρακολουθήσουμε με σωστό τρόπο και την κατάσταση στις υπόλοιπες χώρες. Έχουμε μέσα Μπορούμε να προσκαλέσουμε υπουργού και από την Ελλάδα Θα ακούσουμε από την Επίτροπο τώρα ότι είναι έτοιμη να αναφέρεται σε εμά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα θέματα εφαρμογής των μέτρων που θα αποφουσίσουμε και αυτός είναι ένας ρόλος για μας νομίζω σημαντικός. Πρώτον λοιπόν θα επιταχύνουμε όσο μπορούμε περισσότερο την διαδικασία και δεύτερον θα ελέγξουμε την αποτελεσματικότητα της ίδιας διαδικασίας. Αυτό είχα να πω ως πρόεδρος. Σας ευχαριστώ όλους για τη συζήτηση που προηγήθηκε και θα δώσω το λόγο στην Επίτροπο να δώσει απαντήσεις, πολλές απαντήσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε και σας ευχαριστώ όλους ε, για αυτήν την ε, πολύ επικοδομητική και χρήσιμη συζήτηση. Ε, θα προσπαθήσω να απαντήσω λιγότερο περισσότερο σε όλα τα ερωτήματα ή τα ζητήματα που θέσατε. Ε, καταρχήν σας ευχαριστώ που θέσατε ε, καταρχήν αυτό το ζήτημα προς συζήτηση σήμερα, γιατί είναι αποφασιστική σημασία όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη. Έχετε δίκιο σε αυτό που είπατε, ότι ο, ο στόχος μας είναι βέβαια να φτάσει ο αντίκτυπος στην πραγματική οικονομία, δηλαδή στους δικαιούχους εκείνους που πρέπει να πάνε αυτά τα χρήματα. Και ε, οι, οι ελληνικές υπηρεσίες υιοθέτησαν αυτόν τον μηχανισμό ring fencing, ε, ένα είδος αμυντικού μηχανισμού και μας είπαν ε, δεσμεύθηκαν ότι πράγματι αυτά τα ε, χρήματα θα αξιοποιηθούν μόνο από τους δικαιούχους τους. Ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την πλευρά της θα διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε νέα πληρωμή από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση πράγματι θα φτάσει ε, στου δικαιούχου, δηλαδή θα αποβεί προ όφελο ε, ε, όλα αυτά τα κονδύλια θα αποβούν προ όφελο του ελληνικού λαού. Εγώ βέβαια όπω γνωρίζετε είχα ασκήσει τα καθήκοντά μου σε βουλευτή για 8 χρόνια και πάντοτε ήμουνα υπέρ τη υποστήριξη τη διαδικασία εκείνη η οποία θα ήταν οι καταλληλότεροι, ε, όπου υπάρχει και συζήτηση, αλλά εδώ, όπως αναφέρθηκε ήδη, έχουμε μια εξαιρετική ε, περίπτωση και δεν έχουμε καμία άλλη χώρα η οποία να αντιμετωπίζει ε, μια ίδια κατάσταση δημοσιονομική όπως η Ελλάδα. Οπότε, απαντώντας σε αυτό που είπε ο κύριος Βανίστελροι, έχουμε αυτόν τον ειδικό μηχανισμό τον οποίο εφαρμόζουν οι ελληνικές αρχές και θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτά τα συμπληρωματικά κονδύλια πράγματι θα φτάσουν στην πραγματική οικονομία στους πραγματικούς ε, δικαιούχους. Ε, εγώ προφανώς θα κρατώ ενήμερη ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρέτζη σε ό,τι αφορά την εφαρμογή αυτού του μηχανισμού στο πλαίσιο της, των, της μελλοντικής μας με την Επιτροπή Ρέτζη. Από εκεί και μετά τέθηκαν διάφορα ερωτήματα σε ό,τι αφορά το μνημόνιο και την Τρόικα. Θα ήθελα να πω ευθύ εξ αρχή ότι δεν υπάρχει καμία σχέση ε, μεταξύ αυτών των στοιχείων και ε, του μηχανισμού των διαθροτικών ε, ταμείων. Εμεί ουσιαστικά προσπαθούμε να διαθέσουμε περισσότερα κονδύλια, ώστε να έχουμε περισσότερο βιωσιμότητα και διαθροτικέ μεταρρυθμίσει και προκειμένου να δώσουμε το έναυσμα για περισσότερε επενδύσει στην Ελλάδα. Ελπίζω να απάντησα στα ερωτήματά σας. Ευχαριστώ για την υποστήριξή σας. Η κυρία Κρέλ αναφέρθηκε στο ζήτημα της, ε, του επίγοντος χαρακτήρα και το πόσο σημαντικό είναι να ε, ε, κινηθούμε ταχύτατα και για την περίοδο του 2007-2013 πράγματι είναι πολύ σημαντικό να υιοθετηθούν, να ληφθούν σχετικές αποφάσεις μέσω της επίγουσας διαδικασίας. Γιατί ε, έχουμε αυτό το, την, μικρή δυνατότητα που μας δίνεται, αυτό το παραθυράκι για αυτήν την περίοδο του 2007-2013 ε, καθώς αυτή η περίοδος ε, τελειώνει το Δεκέμβριο του 2015. Και μιλώντας δηλαδή για τον Οκτώβριο είμαστε ήδη καθυστερημένοι, αλλά πραγματικά θα μπορέσουμε να έχουμε ένα θετικό αντίκτυπο αν κινηθούν αντίστοιχα γρήγορα και ελληνικές αρχές. Ε, και κανεί θα αναφέρει το σύστημα των επιπτώσεων. Οι επιπτώσει του να μην υιοθετηθούν αυτά τα μέτρα που προτείνουμε τώρα θα είναι πάρα πολύ σημαντικέ. Καταρχήν η Ελλάδα θα χάσει πάρα πολλά χρήματα. Και από εκεί και μετά, όχι μόνο αυτό, αλλά θα είναι αναγκασμένη η Ελλάδα να επιστρέψει για κάποια κονδύλια. Για να σα δώσω ένα ε, παράδειγμα. Ε, έχουμε ένα αυτοκινητόδρομο ο οποίο έχει ολοκληρωθεί κατά 95%. Εάν δεν ε, ε, δεν υπάρχει σχηματοδότηση για το 5% και αν δεν έχει ολοκληρωθεί αυτό το έργο μέχρι το Δεκέμβριο του 2015 θα πρέπει να επιστραφούν κάποια κονδύλια στην Επιτροπή. Οπότε ε, θα τεθεί κατά κάποιο τρόπο σε κίνδυνο και η νέα προγραμματική περίοδος. Οπότε πραγματικά εδώ μιλάμε για μια ταχεία ενίσχυση ρευστότητας της Ελλάδας ε, και προκειμένου βέβαια το, να αποφευθεί η ε, πιθανότητα να μην υπάρχει ιδιαίτερη εμπιστοσύνη σε ελληνικές ε, τη νέα περίοδο. Προσπαθούμε λοιπόν εδώ να φτάσουμε στην πραγματική οικονομία. Θα ήθελα να απαντήσω πολύ γρήγορα και σε κάποια ακόμα ερωτήματα σε ό,τι αφορά τη διάσκεψη κορυφής του Ιουλίου ε, προφανώς εδώ τα 35 δις που προτείνουμε είναι ε, συμπληρωματικά ε, προς αυτές τις επιστώσεις οι οποίες παραχωρήθηκαν στο πλαίσιο αυτής της διάσημης κορυφής στην Ελλάδα και ελπίζουμε πως όλα, όλες αυτές οι ενισχύσεις από κοινού και στο πλαίσιο του προγράμματος για τη σταθερότητα και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού σταθερότητα θα, φτάσουν, ε, θα έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ε, αυτά λοιπόν τα 35 δις ήδη ε, προβλέπονται ε, στο νέο πολιτικές δημοσιονομικό πλαίσιο. Τα 20 από εκεί προέρχονται από διάφορα διαστατικά ταμεία, ταμείο συνοχής και την πρωτοβουλία για την δημιουργία θέσεων εργασίας και έχουμε άλλα 15 ε, ε, δις τα οποία είναι άμεσες πληρωμές τους ε, Έλληνες γεωργούς μέσω του Ταμείου Γεωργίας και από εκεί και μετά κάποιες πληρωμές από το Ταμείο Αλληλεγγύης. Άρα λοιπόν όλες αυτές οι πιστώσεις εντάσσονται μέσα στο πλαίσιο του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Απλώς προσπαθούμε κάποια από αυτά τα κονδύλια να τα καταβάλουμε ταχύτερα από ό,τι θα συνέβαινε σε μια κανονική περίπτωση. Ε, ευχαριστώ όλους όσους ε, υπογράμμισαν ε, το, το, το ζήτημα του, της, του επίγοντος χαρακτήρα της κατάστασης γιατί πράγματι αν δεν λάβουμε τα μέτρα που προτείνουμε δεν θα είναι σε θέση η Ελλάδα να αξιοποιήσει στο ακέρο όλες αυτές τις επιστώσεις και θέλουμε να μπορέσει η Ελλάδα να αξιοποιήσει γρήγορα αυτά τα κονδύλια ώστε να υποστηρίξει την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και νομίζω πως ε, είπατε επανειλημμένα πως θα πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη σε τέτοιες δύσκολες περιόδους και θα πρέπει να βοηθήσουμε εδώ την Ελλάδα να ενισχύσει την οικονομία της ε, και νομίζω πως ήταν και συναισθηματικά φορτισμένες κάποιες από τις παρεμβάσεις εδώ ε, των μελών της Επιτροπής. Εδώ να πω ότι δεν είναι μόνη χώρα η Ελλάδα που αντιμετωπίζει τέτοιου είδου ε, προβλήματα και είπα στην αρχική μου παρέμβαση ότι θα πρέπει να σκεφτούμε, να κάνουμε κάποιε σκέψει ε, για όλε εκείνε τι χώρε που ε, αντιμετωπίζουν προβλήματα σε ό,τι αφορά την απορρόφηση των κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων και μία από τι προτεραιότητέ μου στο πλαίσιο των νέων μου καθηκόντων είναι ακριβώ να βελτιωθεί η απορρόφηση. Έχουμε 8 χώρε οι οποίε δεν θα μπορέσουν να απορροφήσουν όλα τα κονδύλια από την περίοδο του 2007-2013 όμως η Ελλάδα δεν βρισκόταν σε αυτά, δεν συγκαταλεγόταν σε αυτές τις ε, χώρες ε, τον ε, περασμένο Νοέμβριο, όταν δηλαδή δημιουργήθηκε εκείνο ο μηχανισμός για την βελτίωση της απόρρευσης. Η Ελλάδα δηλαδή βρισκόταν στο 95% πέρυσι τον Νοέμβριο, σε ό,τι αφορά δηλαδή το ποσοστό απορρόφησης των σχετικών κοντιλίων. Και τώρα είμαστε ουσιαστικά στο ίδιο ποσοστό. Δηλαδή δεν ε, συγκαταλεγόταν από την αρχή η Ελλάδα ε, σε αυτόν τον μηχανισμό για την καλύτερη απορρόφηση. Αλλά τώρα αν δεν κάνουμε κάτι θα χαθούν όλα τα υπόλοιπα κονδύλια αν δεν ληφθούν αυτά τα εξαιρετικά μέτρα. Συμφωνώ πάντως ε, με, όλους, με όλα αυτά όσα υπόθηκαν από την κυρία Μάτου, την κυρία Σπυράκη, και άλλος ότι θα πρέπει δηλαδή να εξετάσουμε και την περίπτωση και άλλων κρατωμένων. Αυτό που εγώ προτείνω εδώ και στο πλαίσιο αυτής της συνεδρίασης είναι να βοηθήσουμε την ελληνική οικονομία και να, τις, να παράσουμε μια στρατηγική για να εξέλθει από την κρίση. Και για κάτι τέτοιο χρειαζόμαστε και ένα ε, επενδυτικό σχέδιο, τόσο ώστε τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορέσουν να αξιοποιηθούν ε, Και έχουν δράσει ως σε αυτά τα ταμεία. Όπως γνωρίζετε στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της κρίσης η συμμετοχή ε, σε αυτά τα ταμεία βρισκόταν κατά 35%, ε, ε, κατά 35 υψηλότερο επίπεδο από ό,τι στα εθνικά αντίστοιχα προγράμματα. Οπότε νομίζω πως σωματικά βοήθησαν και στο να αμβληθούν λίγο πτώσεις της κρίσης στην Ελλάδα ήδη από την αρχή αυτά τα ταμεία. Μετά από τα τέσσερα λοιπόν χρόνια συμμετοχή ως κράτος μέλος της Ελλάδας και μετά από 73 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσει στην Ελλάδα έχουμε άλλα 20 δισεκατομμύρια στη διάθεσή μας ε, και εδώ δεν αναφέρομαι ε, μόνο στα διευθυντικά ταμεία. 73 δις λοιπόν έως την ε, προσχώρηση της Ελλάδας. Οπότε Τώρα πρέπει να βασιστούμε και στο τι θα κάνουν οι ελληνικέ αρχέ. Ε, δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα δηλαδή στο πλαίσιο τη επόμενη προγραμματική ε, περίοδου, αλλά έχουμε τώρα τι τροποποιήσεις που θέλουμε να κάνουμε στον κανονισμό με τον... και θα πρέπει βέβαια να γίνονται σεβαστέ αυτέ από όλα τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά επενδύσει ε, στου κύριου τομεί που περιλαμβάνονται και στην ε, στρατηγική 2020, έρευνα και καινοτομία, ε, ενέργεια, αστική ανάπτυξη, ε, κοινωνική ένταξη και ούτω καθεξής. Είναι λοιπόν αρμόδιες οι ελληνικές αρχές για να υλοποιήσουν αυτή τη στρατηγική στην πράξη, να δώσουν δηλαδή τις προτεραιότητες, να εντοπίσουν και να υλοποιήσουν τα προγράμματα εκείνα που είναι απαραίτητα και είναι υψηλής ποιότητας. Ε, όπως όμως είπα, 35 χρόνια λοιπόν εμπειρία σε ό,τι αφορά την υλοποίηση τέτοιων ε, ε, ταμείων και νομίζω πως όλοι όσοι έχουν επισκεφθεί την Ελλάδα ε, μπορούν να διαπιστώσουν τις αλλαγές που έχουν γίνει, τις πραγματικές αλλαγές που έχουν επέλθει στην Ελλάδα. Εγώ κάτι την τετραήμερη μου επίσκεψη στην Ελλάδα είχα εκπλαγεί από το γεγονός ότι συχνά δεν αναφερόμαστε σε όσα καταφέρνουμε να κάνουμε στα κράτη-μέλη και τη διαφορά την οποία τελικά κάνουμε. Δηλαδή, αν κάποιο πήγαινε στη δεκαετία του 80 στην Ελλάδα και έκανε, έβγαζε κάποιε φωτογραφίε και την εμπιστευτόταν τώρα, θα, ε, ότι βρίσκεται σε έναν άλλον αιώνα. Δηλαδή, πραγματικά θα πρέπει να είμαστε περήφανοι με αυτά που έχουμε καταφέρει και μέσω των διαρθωτικών ταμείων, όχι μόνο βέβαια στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλα κράτη-μέλη. Και να σα δώσω κάποια παραδείγματα. Ε, για παράδειγμα ε, σύνδεση της υπηρετικής Ελλάδας με την ε, Πελοπόννησο, μια πολύ μεγάλη γέφυρα, κύριο, δηλαδή, κάποια πολύ μεγάλα νοσοκομεία τα οποία συγχρηματοδοτήθηκαν, το μετρό των Αθηνών, νέα σχολεία και μιλάμε για δεκάδες Αθηναίων οι, οποία, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιούν αυτό το ε, δίκτυο του μετρό έχουν επενδυθεί 5 δισεκατομμύρια ευρώ ε, ε, σε αυτό το, στο δίκτυο του μετρό και στο πλαίσιο μια συνέντευξη σήμερα είναι ένα δημοσιογράφο ε, μου είπε εκείνο ότι υπήρξαν κάποια κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ήταν κάποια. Υπήρξαν πάρα πολλά δισεκατομμύρια που έχουν πραγματικά επιφέρει αλλαγέ. Είχαμε ε, δώσει και βοήθεια κατά τη διάρκεια των ε, πλημμύρων σε ό,τι αφορά για παράδειγμα και άλλε προγράμματα διαχείριση αποπλήτων και λιμάτων. Και εδώ αναφέρω για παράδειγμα όλα αυτά τα προγράμματα ενδεικτικά με τα οποία έχουμε βοηθήσει την Ελλάδα. Νομίζω πως θα πρέπει να γίνει και ε, μια περαιτέρω συζήτηση ε, με την Επιτροπή σας σε ό,τι αφορά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και άλλα κράτη-μέλη, αλλά πραγματικά εδώ στην περίπτωση της Ελλάδας έχουμε να κάνουμε μια ειδική περίπτωση. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία άλλη χώρα που να αντιμετωπίσει τα, την ίδια κατάσταση σε επίπεδο δημοσιονομικό με την Ελλάδα. Και ακριβώς τα μέτρα που προσπαθούμε να λάβουμε απευθύνονται στην αντιμετώπιση αυτής της ε, κατάστασης. Δηλαδή διάθεση κατάλληλη ρευστότητας και υλοποίηση επενδύσεων ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στην πραγματική οικονομία. Αλλά ε, συμφωνώ με τον κύριο Πετσολίνο και όλους όσους είπαν ότι ε, χρειάζεται πράγματι να γίνει μια γενικότερη συζήτηση, δηλαδή σε ό,τι αφορά και όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Θα σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτή τη συζήτηση. Ε, σε ό,τι αφορά την τεχνική αρρωγή, να πω ότι σας διαβεβαιώ ότι οι υπηρεσίες της ελληνική ε, Διεύθυνσης ε, Ρέτζιο συνεργάζονται στενά με τις ελληνικές υπηρεσίες τους ώστε να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά τα καμπτήλια. Κάποιοι εμπειρογνώμονες ε, από την Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο ήδη έχουν αποσπαστεί στο Υπουργείο Οικονομικών ώστε να βοηθήσουν στο σχεδιασμό των νέων project και να απαντήσουν κάποια ερωτήματα σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την, τους διαγωνισμού. Ε, το σχέδιο Juncker και άλλα ζητήματα τα οποία χρειάζονται διευκρινήσεις. Ε, πάντως ε, πράγματι συμφωνώ με αυτό που υπόθηκε ότι δηλαδή και οι διοικητικές δυνατότητες μερικές φορές είναι πολύ σημαντικές, σημαντικότερες και από τα ίδια τα χρήματα και είναι σημαντικό δηλαδή αυτές οι δυνατότητες διοικητικές να επεκταθούν και να βελτιωθούν σε πολλές χώρες ούτως ώστε για παράδειγμα να είναι πιο ανθεκτικέ και στη διαφθορά, πιο ανθεκτικέ στην απάτη, να υπάρχει ένα καλύτερο σύστημα ελέγχων στο πλαίσιο των ε, διοικήσεων και μέσω της κοινή ομάδα εργασία ε, την οποία έχουμε δημιουργήσει προσπαθούμε ακριβώς να ε, ασχοληθούμε με αυτά τα ζητήματα. Κοινή ομάδα εργασία δηλαδή μεταξύ ελληνικών αρχών και επιτροπή και υπάρχει και μια ε, νέα ε, υπηρεσία υποστήριξη των διαφθορτικών μεταρρυθμίσεων η οποία θα αποτελεί ακριβώς ένα ακόμα κανάλι αν θέλετε για την διαβίωση νομοσύνης προς την Ελλάδα. Ε, ο στόχος μας λοιπόν είναι να επιταχύνουμε την υλοποίηση των σχετικών προγραμμάτων, να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών στην Ελλάδα και όταν μιλάμε για το επίπεδο της ε, εφαρμογής, πάντα βέβαια εκεί έχουμε να κάνουμε και με την ευθύνη των ίδιων των κρατών πώς θα προχωρήσουν δηλαδή με την υλοποίηση των επενδύσεων. Εμείς ε, προσπαθούμε λοιπόν να βοηθήσουμε όπως μπορούμε με μια τέτοια ταχεία ένεση ρευστότητας και η Ε, από εκεί και μετά, ε, σε ό,τι αφορά την επίγουσα διαδικασία, αυτό θα εξαρτηθεί από την απόφαση που θα λάβετε εσείς από κοινού Κοινοβούλιο και Συμβούλιο. Σε ό,τι αφορά τώρα την ανθρωπιστική κρίση θα ήθελα να πω δύο λόγια. Γνωρίζουμε ε, πολύ καλά ότι έχουμε πολύ λεπτές και δύσκολες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σε αυτό το επίπεδο και η πολιτική συνοχή έχει ήδη ε, συμβάλλει στην κοινωνική ένταξη των μεταναστών ε, σε πολλά σημεία ε, και δεν αναφέρουμε μόνο στις χώρες οι οποίες πλήγονται ιδιαίτερα τώρα τελευταία αλλά αναφέρουμε για παράδειγμα σε προάστια του Βερολίνου, του Παρισίου και είδα εκεί ότι υπάρχουν πράγματι υλοποιούνται ε, μία σειρά από προγράμματα για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών. Και θα ήθελα ε, να σας διαβεβαιώσω ότι από την πρώτη μέρα που επέστρεψα από το καλοκαιρινό ε, διάλειμμα κάναμε μία εκτεταμένη συζήτηση εντός της Γενικής Διεύθυνσης Ρίτζιο και προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να δώσουμε, να παράσουμε περαιτέρω βοήθεια ούτως ώστε να κάνουμε κάποια μεταβίβαση σε ό,τι αφορά κάποια μετάθεση των ε, προτεραιοτήτων, ούτως ώστε για παράδειγμα να δώσουμε τη δυνατότητα για υποστήριξη σε ό,τι αφορά ε, καταλήματα, ψυχολογική υποστήριξη, ειδικότερα σε συνοριακά σημεία διέλευσης ε, και το πώ μπορούμε να διέσουμε και σχετικά κονδύλια για την περίοδο 2014-2020 νομίζω πως η λέξη κλειδί θα είναι η ένταξη, το integration και νομίζω πως κάποια κράτη-μέλη ήδη έχουν αξιοποιήσει τέτοια κονδύλια όπως για παράδειγμα η Ιταλία. Η Ιταλία αξιοποίησε ε, στο πλαίσιο του προγράμματος Σικουρέτσα ε, ε, όλα τα κονδύλια της περίοδου 2007-2013 δημιουργώντας 100 ε, σημεία καταλήμματων για ε, τις ε, περιοχές οι οποίες είχαν πληγεί περισσότερο όπως η Απούλια, Κατάνια και άλλες και δεν λέμε ότι θα, κάνουμε, θα έχουμε περαιτέρω γενικότερη ε, ανακατανομή ε, ούτως ώστε να διατεθούν περισσότερα ε, κονδύλια για τη μετανάστευση αλλά το κάθε κράτος μέλος μπορεί να, θέσει, να κάνει έτοιμα ούτως ώστε να λάβει μια περισσότερη βοήθεια και έχουμε καλά παραδείγματα από το παρελθόν για παράδειγμα στις κάτω χώρες υπήρξε μια γυναίκα από την Ιορδανία είχε την ιδέα να διαθέτει κάποια προϊόντα της Ιορδανίας στην αγορά εκεί ε, και έχει για παράδειγμα δημιουργήσει μια οικογενειακή επιχείρηση που την βοηθάει και έχουμε για παράδειγμα δημιουργήσει τέτοιους μηχανισμούς σε διάφορες χώρες για startups, ε, δηλαδή για μικροεπιχειρήσεις. Γιατί μιλάμε βέβαια πολύ συχνά για μετανάστες οι οποίοι έχουν πολύ ε, καλές δεξιότητες, μιλάμε δηλαδή για γιατρούς ε, και άλλους υψηλά ανθρώπους, οπότε θα πρέπει να ε, διαθέσουμε και εμείς τα απαραίτητα κονδύλια τους ώστε να μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε νομίζω εξαντλήσει, δεν έχουμε ψάξει σωστά και με το Interreg και τα άλλα προγράμματα τα διαμεθοριακά νομίζω ότι ίσως ε, δύο εβδομάδες μετά το Στρασβούργο κάποιοι από εσά θα βρεθείτε στο Λουξεμβούργο για να γιορτάσουμε τα 25 χρόνια των προγραμμάτων Interreg. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού όλα αυτά τα προγράμματα τα οποία βρίσκονται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφησαν όπως επίσης και αυτά τα οποία ισχύουν με χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Σερβία, ε, τέος Γιουκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, και θα πρέπει να δούμε αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιες από τις πιστώσεις αυτές στη σημερινή συγκυρία και για τη διευκόλυνση των μεταναστών. Λοιπόν, ε, σας ευχαριστώ για τη συνάντηση αυτή. Θα συναντηθούμε στην Ολομέλεια την επόμενη εβδομάδα και με χαρά θα συνεργαστώ για μια ακόμη φορά μαζί σας. Όπως σας υποσχέθηκα, ε, θα επανέλθουμε για να σας δείξουμε πώς θα εφαρμοστούν τα μέτρα αυτά, όχι μόνο για την Ελλάδα. Ξέρετε ότι το 2016 είναι ένα κρίσιμο έτος για όλους. Είναι το πρώτο έτος όπου θα δούμε πλέον απτά αποτελέσματα του τρόπου με τον οποίο διαφοροποιούν την κατάσταση επιτόπου οι παρεμβάσεις μας. Thank very much, Σας ευχαριστώ Επίτροπε. Λοιπόν, όλες σχεδόν οι ερωτήσεις βρήκαν τις απαντήσεις τους. Λοιπόν, αυτά. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Ο κύριος Βανίστελόι. Ευχαριστώ πολύ. Η συνάντηση αυτή ήταν κάτι το οποίο αφορούσε κυρίως τη διαδικασία. Ας προσπαθήσουμε να καταλήξουμε κάπου σε επίπεδο διαδικασίας. Εγώ είπα ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα προτιμά την κανονική διαδικασία. Λόγω όμως της συγκυρίας, λόγω του ότι εμείς θα πρέπει να δούμε το τι θέλουμε να κάνουμε σαν κοινοβούλιο. Άκουσα τα σχόλια κάποιων από τον συναδέλφο και μου έκαναν εντύπωση. Είναι σαφές ότι εμείς θα στηρίξουμε το πακέτο αυτό για την Ελλάδα και την προχρηματοδότηση και τις επενδύσεις λοιπά. Αλλά αν δεν εμείνουμε στο ρόλο μας, γιατί να μην έχουμε ένα ειδικό εισηγητή για το 16 στην Επιτροπή μας για την Ελλάδα. Ξέρουμε, λέμε γενικά ότι οι επενδύσεις θα πρέπει να πηγαίνουν ε, απευθείας εκεί που πρέπει, σε αυτούς οι οποίοι θα πρέπει να ε, ωφεληθούν συνένα και τα λοιπά σαν κοινοβούλιο εν πάση περιπτώσει εμείς θα πρέπει να έχουμε κάποιον ο οποίος να παρακολουθεί από κοντά τις υποθέσεις αυτές και να ενημερώνει τις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Εσείς θα κάνετε μια συγκεκριμένη διαδικασία επί του διαδικαστικού, μια συγκεκριμένη πρόταση επί του διαδικαστικού, δεν ξέρω, με μια επιστολή, με κάποιο τρόπο θα εκφάσετε την άποψη της Επιτροπής μας. Δεν μπορούμε να πούμε απλά ότι «Α, εντάξει, ερωτήθηκε το Κοινοβούλιο και είπε ναι στη διαδικασία η οποία προτείνεται». Όχι. Υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία τα οποία μας απασχολούν και θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι για το 2016 μπορεί να χρειαστεί να γίνουν κάποιες συναλλικότερες συζητήσεις να πάρουμε εμείς την πρωτοβουλία για τις ε, εξελίξεις και να μην περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε φορά που έχει μια δυσκολία να προσφέρει σε εμάς σε βιαστική. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτή την έκτακτη κατάσταση Ίσως όμως να χρειάζονται και κάποιες περισσότερες ενέργειες από πλευράς μας για να λειτουργήσουμε πιο, ε, θα έλεγα, πιο προβλεπτικά. Θα υποστηρίξω λοιπόν τη μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων και όπως είπα θα πρέπει να δούμε τι γίνεται στο Συμβούλιο. Γιατί αν τώρα κατέβει το Συμβούλιο ξαφνικά και καταθέσει τροπολογίες, ε, τότε υποχρεωτικά εμείς δεν θα καταπιούμε τις τροπολογίες αυτές αμάσιτες, θα πρέπει να τις επανεξετάσουμε, θα πρέπει να τις συζητήσουμε. Λοιπόν, εγώ αρχικά πίστευα ότι πρέπει να ακολουθήσουμε την τακτική διαδικασία, με έκτακτες συνεδριάσεις για να μην χαθεί χρόνος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η πλειοψηφία αποφασίζει διαφορετικά. Θα στηρίξουμε την απόφαση αυτή, αλλά όμως η Επιτροπή μας να είναι διαθέσιμη να πάρει την πρωτοβουλία. Όπως ε, επισήμανα και στην αρχή, η Επιτροπή και για την περίπτωση της Ελλάδας και των άλλων χωρών που είναι σε πρόγραμμα άργησε να πάρει πρωτοβουλίες προκειμένου να υπάρχει μια σημαντική απορρόφηση άμεση τις παρατηρήσεις μου για το ρόλο του μνημονίου στην Ελλάδα και το πρόγραμμα το καινούργιο τις έκανα. Αυτό δεν πρέπει να το συγχαίουμε με τα μέτρα που πρέπει να πάρουμε τώρα και κατά την έννοια αυτή εμείς από την αρχή και το είπα είμαστε υπέρ της διαδικασίας που είναι ταχύτατη. Έχουμε μια έκτακτη διαδικασία επομένως πρέπει να πάμε σε αυτόν τον κανονισμό που προτείνεται ως μια διαδικασία άμεση η οποία μπορεί να ξεμπλοκάρει και να δώσει την ευκαιρία παρά τα λάθη που έγιναν και από την Τρόικα και στην Ελλάδα και τα προβλήματα που υπάρχουν παρόλα αυτά σήμερα χρειαζόμαστε άμεση δράση. Το έχω πει πολλές φορές στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε εσά κυρία Επίτροπε για το ποια άμεσα μέτρα θα πρέπει να πάρουμε. Επομένως πρέπει να πάμε με την απλουστευμένη διαδικασία κύριε συνάδελφοι του Λαϊκού Κόμματος ξεκάθαρα να περάσει αυτή η διαδικασία να προχωρήσει και φυσικά τόσο οι δικές μας παρατηρήσεις όσο και άλλες παρατηρήσεις να ληφθούν υπόψη διότι θα πρέπει να ανοίξει ένας σοβαρός διάλογος. Είναι σίγουρο ότι χρειάζεται αλλαγή και το σύμφωνο σταθερότητας και οι επενδύσεις να μην μετράνε στο έλλειμμα και οι χώρες που βρίσκονται υπό εποπτεία να μπορούν να κάνουν επενδύσεις και να μην μπαίνουν στη διαδικασία του περιορισμού των ελλημάτων. Αυτά είναι θέματα που πρέπει να τα δούμε όπως και την απορρόφηση. Ξεκάθαρα πρέπει να τα πάμε έτσι. δεν συμφωνώ με ένα ειδικό ραπορτέρ για την ελλάδα που θα μπει υπό την εποπτεία του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου. πιστεύω ότι όλα πρέπει να είναι ανοιχτά σε ισότιμη βάση να ελέγχουμε όλε τι χώρε, αλλά εδώ έχουμε έκτακτε καταστάσει, χρειαζόμαστε έκτακτε αποφάσει, επομένω με την απλουστευμένη διαδικασία να προχωρήσουμε. είναι ξεκάθαρο το είπα από την αρχή ότι άργησε η επιτροπή να προχωρήσει σε αυτή την κατεύθυνση. ευχαριστώ. Thank you. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Νοβάκοφ ζήτησε 30 δευτερόλεπτα χρόνο. Παρότι δεν είμαι ειδικό. Ε, ξέρω ότι υπάρχουν ε, προβλήματα με όλε τι χώρε που ε, πρέπει να εφαρμόσουν αυτά τα διαρθρωτικά προβλήματα. Χρειαζόμαστε απλούστευση, διότι οι κανονικέ διαδικασίε είναι πολύ ταχείε και ταυτόχρονα χρειάζονται πάρα πολλά έγγραφα και είναι πολύ χρονοβόρε. Γι' αυτό σα ζητώ. Κυρία Επίτροπε, να κάνετε ό,τι μπορείτε για να επιταχύνετε τη διαδικασία απλούστευσης στην πολιτική συνοχής διότι ε, πρέπει να περιορίσουμε τη γραφειοκρατία το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστώ. Κυρία Κχέλ, που θα είναι και η τελευταία παρέμβαση. Θα είμαι πολύ σύντομη και εγώ, λέει η κυρία Κχέλ. Βλέπω ότι από τη σημερινή συζήτηση προκύπτει ότι όλες οι πολιτικές ομάδες συμφώνησαν ότι θα εφαρμόσουμε την απλουστευμένη διαδικασία. Και θα ήθελα να ακολουθήσουμε την πρόταση του κυρίου Βανίστερ Ρόι στην επόμενη συνάντηση συντονιστών να συζητήσουμε τι μπορούμε να κάνουμε σε πλαίσια αυτή τη απλουστευμένη διαδικασία για να παρακολουθούμε την όλη αυτή διαδικασία. Ελπίζω ότι αυτό θα είναι το αποτέλεσμα και η διαπίστωση αυτή τη συνάντηση για να συνεχίσουμε τις εργασίες μα. Ευχαριστώ. Καλώς, ευχαριστώ πολύ λέει η Πρόεδρος. Ναι, ακριβώς περί αυτού πρόκειται. Μετά από όλε τις συζητήσεις που έγιναν, ως πρόεδρος προτείνω να λάβουμε μια απόφαση υπέρ της απλουστευμένης διαδικασίας. Σύμφωνα με το άρθρο 50 του κανονισμού του Κοινοβουλίου, το σημείο 1 του άρθρου 50, ε, όπου λέει τα εξής μετά την πρώτη συζήτηση για μια πρόταση νομοθετικής πράξης, ο πρόεδρος μπορεί να προτείνει έγκριση χωρίς τροπολογίες. Αυτό ακριβώς το οποίο σας προτείνω λοιπόν. Εκτός εάν ένα δέκατο των μελών της Επιτροπής έχουν αντίρρηση. Αν δεν έχουν αντίρρηση το ένα δέκατο των μελών, ε, ο πρόεδρος υποβάλλει στο Κοινοβούλιο μια έκθεση για έγκριση της διαδικασίας άρθρο 151, δεύτερη υποπαράγραφος 2 και 4. Το 1 δέκατο της Επιτροπής μας σημαίνει 5 μέλη της Επιτροπής. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν αν υπάρχει κάποιος που έχει αντίρρηση με την απλουστευμένη διαδικασία. να ψηφίσουμε σημαίνει κάτι άλλο, λέει ο κύριο Βανίστερόι. Ναι, εγώ θέλω να ρωτήσω αν έχει κάνει αντίρρηση, λέει η πρόεδρος. Και από ό,τι βλέπω κανείς δεν έχει αντίρρηση. Μία αποχή μόνο. Μία αποχή. Θα θέλαμε πέντε διαφωνούντες και έχουμε μία αποχή μόνο. Να ψηφίσουμε ή δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε. Θα υποβάλω λοιπόν την έκθεσή μας. Συμφωνούμε λοιπόν ότι είναι σαφής η διαδικασία που ακολουθούμε. Ωραία, συμφωνούν όλοι λοιπόν με τη διαδικασία αυτή που ακολουθούμε. Μπράβο μας. Okay. Thank you everybody. Thank you. Σας ευχαριστώ όλους. Σας ευχαριστώ για τις ιδιαίτερα επικοδομητικές σημερινές συζητήσεις και σας εύχομαι καλή σύνοδο την επόμενη εβδομάδα και θα το πούμε στις 17.